Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με μεγάλη χαρά και αισθανόμενη ειλικρινή τιμή, μία κοινοβουλευτική επιτροπή, η δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή, και θα έλεγα και το Ευρωκοινοβούλιο το ίδιο οργανώνει αυτή την εκδήλωση για τους πολίτες, Citizens Event, και με τους συναδέλφους βουλευτές που βρίσκονται στην αίθουσα, θα εγκαινιάσουμε αυτήν την εκδήλωση. Ανοίξαμε διάπλατα τις πόρτες του Κοινοβουλίου στους πολίτες, αλλά και τις πόρτες της Επιτροπής μας, της Επιτροπής που ονομάζεται Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ήρθατε σε μεγάλο αριθμό σήμερα, περίπου 150 πολίτες από όλες τις γωνιές της Ευρώπης για να μας μιλήσετε και να μας θέσετε ερωτήσεις. Το επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό για μένα και τους συναδέλφους μας να έχουμε αυτό το διάλογο, τον απευθείας διάλογο μαζί σας και να σας ακούσουμε. Θέλουμε να αφουγκραστούμε τις απόψεις σας, τις επιθυμίες σας, τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ την κυρία Γκραπίνη, η οποία προσκάλεσε μια αντιπροσωπεία από την χώρα της, τη Ρουμανία. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Εκπροσωπούνται κάτω χώρες με τον δικό μας Βιν Βαντεκάμπ, Βεβαίω ο αντιπρόεδρό μα ο κ. Κοκ με μια αντιπροσωπεία από τη Γερμανία. Καλώ ήρθατε κι εσεί. Η Γαλλία επίση εκπροσωπείται με μια ομάδα στο βάθο τη αίθουσα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είστε κι εσεί δεκτή. Η αντιπροσωπεία από τη Γαλλία είναι πολύ σύνθετοι συνδικαλιστές, φοιτητές, πολλοί κόσμος. Δεν θα πω και ονόματα, μην χαμογελάτε ε, ύποπτα συνδικαλιστές και σε αυτή την αίθουσα θελήσαμε να βεβαιωθούμε ότι θα διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση ό,τι και αν γίνει. Γιατί οι μεταφορές είναι η καθημερινότητά μας. Γι' αυτό. Είναι η διαδρομή που κάνετε από το σπίτι στη δουλειά. Οι μεταφορές καθορίζουν το σημείο που θέλουμε να κατοικήσουμε, σε ένα αστικό κέντρο ή στην εξοχή αφορούν την υγεία μας, αφορούν τον αέρα που αναπνέουμε οι μεταφορές. Σε ένα βαθμό καθορίζουν και το πορτοφόλι του καθενός, το προπολογισμό μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 13% του προπολογισμού δαπανάται στις μεταφορές. Κυρίως όμως επειδή τη μεγαλύτερη πρόκληση του αιώνα δεν θα την αντιμετωπίσουμε αν δεν αλλάξουμε του τρόπου μεταφορά μα. Μιλάω για την υποχρέωση όλων μα σε αυτήν την αίθουσα. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο να σώσουμε τον πλανήτη. Προ στιγμή το κλίμα δεν τα πάει καλά. Όταν ε, λέμε μεταφορέ δεν πρέπει να ξεχνάμε την πρόκληση, την πρόκληση των κλιματικών αλλαγών. Έχουμε λοιπόν ηθική υποχρέωση να φέρουμε αποτέλεσμα, να μειώσουμε τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου. Διότι το θυμίζω και αυτό από σήμερα έως το 2050 πρέπει κατά 60% να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Και είναι ένα παράδειγμα μόνο αυτό, γιατί ο τομέας των οραμεταφορών νομίζω προσωπείται σε αυτή την αίθουσα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, θα πρέπει να δουλέψουμε εδώ για τις αερομεταφορές, ο τομέας αυτός μόνο θα τριπλασιάσει τις εκπομπές του το 2000. Θα τριπλασιαστεί μάλλον στον όγκο του το 2050. Πρέπει λοιπόν να μειώσει τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Και κάτι άλλο που είναι επίσης σημαντικό, η ευρωπαϊκή διάσταση. Οι μεταφορές είναι άνοιγμα προς τον άλλον, είναι άνοιγμα για τον άλλον. Είναι κάτι που μας επιτρέπει να ε, ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε αυτό το μεγάλο ανθρώπινο εγχείρημα, το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σε αυτό λοιπόν το σώμα, ε, σε αυτό το κτίριο ερχόμαστε κάθε μέρα με την ελπίδα ότι καθημερινά θα διασυνδέσουμε ακόμη περισσότερο και καλύτερα τους Ευρωπαίους πολίτες μεταξύ τους. Αυτό το πάθος και τον ενθουσιασμό θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας σήμερα. Και πραγματικά ως πρόεδρος θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κάνατε να έρθετε ως εδώ, να είστε μέσα στην αίθουσα και πραγματικά θα χαρούμε που θα σας ακούσουμε. Να σας παρουσιάσω την ομάδα μας για το δύο ώρα που θα ακολουθήσει. Για μένα είναι σημαντικό να αντιληφθείτε ότι χρειάζονται κάποια κλειδιά για να μπορέσετε να ε, αντιληφθείτε τον τρόπο που λειτουργούν ε, τα θεσμικά μας όργανα. Η αίθουσα στην οποία εργάζεστε, όχι δεν εργάζεστε, στην οποία σας υποδεχόμαστε, η αίθουσα αυτή είναι αίθουσα εργασίας. Αίθουσα εργασίας, στην εργασία μας, στην αρμοδιότητά μας ως συνομοθετών. Δηλαδή εδώ συμμετέχουμε στην σύνταξη των νόμων. Οι βουλευτές στις επιτροπές τους συνέρχονται στις συνεδριάσεις ανάλογα με το πολιτικό τους βάρος στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλες μας οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες, ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά. Η διαφάνεια είναι έμφυτη στην ουσία και τη φύση του δημοκρατικού διαλόγου και αυτό επιδιώκουμε και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι συνεδριάσεις μας μεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ένα πολύγλωσσο κοινοβούλιο το οποίο λειτουργεί πολύ καλά χάρη στην πολύ ταλαντούχα ομάδα διερμηνίας που έχουμε μαζί μας και θα σας παρακαλέσω να τους χειροκροτήσετε γιατί θα μείνουν μαζί μας όλο το απόγευμα και ποτέ δεν τους ευχαριστούμε αρκετά. Έχετε μπροστά σας, μεταξύ ε, αγαπητοί μου μάλλον συμπολίτες, ε, αρκετούς ευρωβουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες στο Προεδρείο, πώς οργανωνόμαστε στο Προεδρείο, στο Προεδρείο έχουμε αντιπροέδρους της Επιτροπής. Ο κύριος Κόχ είναι αντιπρόεδρος, ο κύριος Ρικέ που θα φτάσει όπου να είναι, είναι επίσης αντιπρόεδρος και γενικώ είναι αυτοί που είναι αντιπρόεδροι μετά από μένα. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Εντάξει. Έπειτα έχουμε πολύ σημαντικέ προσωπικότητες στην Επιτροπή μας, τους οποίους θα ονομάσουμε συντονιστέ. Οι συντονιστέ είναι βουλευτές κάπω ιδιαίτεροι, διότι έχουν αναλάβει το καθήκον να προσδιορίσουν και να προσανατολίσουν την γραμμή της ομάδας τους, ε, δίνοντας μια κατεύθυνση ε, στις συζητήσεις και την εξέταση των θεμάτων εντός της ομάδας τους. Να τους αναφέρω. Ο κύριος Βιμ Βαντενκάμπ, Κύριε Βαντενκάμπ, μπορείτε να σηκωθείτε. Σηκωθείτε, παρακαλώ. Συντονιστή τη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου. Ο συντονιστή τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριο Ισμαήλ Ερτούγκ. Ο κύριος Ρόμπερτ Ζήλε, ο οποίος είναι συντονιστής των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, εδώ, στην Επιτροπή μας. Ο κύριος Τέλιντσκα, ο οποίος είναι συντονιστής της ομάδας Άλντε των Φιλελευθέρων. Ο συντονιστής των Πρασίπων, Πρασίνων, ο κύριος Νταλούντε, Γιάκομ Νταλούντε. Και πολλοί άλλοι ευρωβουλευτές στην Επιτροπή μας οι οποίοι είναι όλοι ειδικοί ε, επί του θέματος, είναι παίοντες για θέματα μεταφορών και τουρισμού. Τώρα, γιατί επιλέξαμε αυτό το ιδιαίτερο θέμα για τις μεταξύ μας συζητήσεις και το διάλογο. Γιατί πραγματικά σήμερα θέλουμε να επεξεργαστούμε το θέμα του μέλλοντος, το μέλλον των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου θα διοργανώσουμε αυτή τη συζήτηση επί ένα δίωρο ως εξής. Μας παρακολου... Επειδή μας παρακολουθούν τα κοινωνικά δίκτυα, και επειδή μεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίασή μας, θα έχετε ζωντανά τη δυνατότητα να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Απευθείας στους βουλευτές της αρεσκίας σας, αλλά και στους προσκεκλημένους μας. Η ακρόαση, συζήτηση θα οργανωθεί θα διορθωθεί σε δύο τμήματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε προσκαλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα μιλήσει για το μέλλον των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπροσωπείται από τον κύριο Πακέ στα αριστερά μου, ο οποίο είναι αναπληρωτή γενικό γραμματέα και, ε, στην και μάλλον στο ιστορικό του έχει μια μακρά εμπειρία στον τομέα των μεταφορών. Επίσης, μετά θα δώσω το λόγο σε εσά τους πολίτες, όσους είστε εδώ, θα είστε ελεύθεροι να θέσετε ό,τι ερώτηση σας αρέσει. Στους συντονιστές, στους βουλευτές, σε όποιον θέλετε. Και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε και θα επιλέξουμε και κάποιες ερωτήσεις από τα κοινωνικά δίκτυα. Αν κάνετε σχόλια στο Twitter και το καθεξής, το hashtag είναι hashtag ε, μέλλον 4 tran. Future for tran. Και στο δεύτερο μέρος της συζήτησης θα δώσω το λόγο στον Ξαβιέ Τοκέν, ο οποίος έρχεται από την φαμπρίκ της κινητικότητας και θα ξανακούσουμε ερωτήσεις από, την, ε, από το κοινό. Μετά θα κλείσουμε τη συζήτηση κάνοντας μια ανακεφαλαίωση της σημερινής εμπειρίας. Θα ε, δούμε λίγο τους κανόνες. Ε, να πω στους, παρε, στους ε, ότι θα είναι αδιάλακτη. Ο χρόνος ομιλίας θα είναι 10 λεπτά, θα υπάρχει χρονόμετρο, διότι τον λόγο σήμερα θέλει να τον πάρουν οι πολίτες. Και έχετε κι εσείς πολίτες μου υποχρεώσεις όταν παίρνετε το λόγο. Θα μας λέτε από πού έρχεστε και το ονοματεπώνυμό σας να συστήνεστε για να μπορούμε κι εμείς να ξέρουμε ποιον ακούμε. Υπάρχει κάποια ερώτηση περί μεθοδολογίας? Όχι. Να αρχίσω ευθύ αμέσως, δίνοντας λοιπόν το λόγο για 10 λεπτά και θα βάλω το χρονόμετρο αμέσως να τρέχει στον κύριο Ζαν Ερικ Πακέ, ο οποίος είναι απληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο, κύριε Πακέ, αλλά με μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, για την πρόσκληση. Είναι πολύτιμος ο χρόνος στο Ευρωκοινοβούλιο και θα παραμείνω εντός του δεκαλέπτου. Να σας πω ότι ο διάλογος με τους πολίτες που διοργανώνεται από την Επιτροπή Τραν και την Πρόεδρό της σήμερα το απόγευμα εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία. Διαδικασία διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών ε, θεσμικών οργάνων και των αρχών των κρατών μελών των αρχών των κρατών και των περιφερειών. Για το μέλλον των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε το Μάρτιο αυτή τη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλη η πρωτοβουλία και ανέλαβε ένα μεγάλο μέρο τη στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και κυβερνήσει των κρατών μελών. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το συζήτησαν στη σύνοδό του στο Τάλιν πριν από λίγε μέρε και θα συνεχίσουν τι συζητήσει και μεταξύ του διασφαλίζοντας ότι στη συζήτηση με τους όλους πολίτες γίνονται σεβαστές οι αρχές της δημοκρατίας, Σε μια εκδήλωση όπως αυτή που ε, έχετε προσκληθεί σήμερα το απόγευμα. Για να μπορούν οι πολίτες να ε, επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί μας το μέλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει επιλεγεί πολύ εύστοχα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Είναι καθοριστικό το θέμα αυτό. Οι μεταφορές κάνουν την Ευρώπη κάτι χειροπιαστό, μια πραγματικότητα. Η Ευρώπη είναι το πραγματικό σας, το αληθινό σας ενδιέτημα, εκεί που κατοικείτε. Εκεί ζείτε, εκεί φυτάτε, εκεί μετακινήστε για την ψυχαγωγία σας, για να επισκεφτείτε την Ήπειρό μας. Αλλά το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν είναι ένα φυσικό, ε, ένα αθόρμητο εγχείρημα. Είναι κάτι που βασίστηκε σε πολιτικές αποφάσεις. Το σκέφτηκε, το αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι και το πρότειναν. Γι' αυτό βασίζεται στο διάλογο. Στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον ε, της Ευρώπης που συζητιέται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και θα συζητιέται στι ευρωεκλογέ του 2019. Σε αυτό το πλαίσιο οι μεταφορές είναι προφανώς στον πυρήνα του όλου προβληματισμού και είναι ζωτική σημασία γιατί είναι ένα τομέα που τον ζουν οι πολίτε καθημερινά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην άμεση καθημερινότητα. Γι' αυτό ο διάλογο σήμερα πιστεύω πρέπει να ασχοληθεί με το περιεχόμενο των ευρωπαϊκών πολιτικών αλλά πρέπει να ενσκύψει και στο καλύτερο δυνατό τρόπο διάρθρωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών μεταξύ τους σε θέματα μεταφορών ποια είναι η θεώρησή μας για το μέλλον των ε, πολιτικών μεταφοράς στην Ευρώπη. Τι θα γίνει σε εθνικό επίπεδο, τι θα κάνουν οι περιφέρειες, οι δημοτικές αρχές, αλλά και τι θα υλοποιηθεί σε ακόμη τοπικότερο επίπεδο, στα αστικά κέντρα. Η δουλειά αυτή, η προσπάθεια διάρθρωσης πρέπει να γίνει όχι μόνο σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, αλλά και τον αρμόδιο βιομηχανικό κλάδο των μεταφορών. Ο τομέα των μεταφορών είναι ένα από του πλέον ενδιαφέροντε τομεί και απεικονίζει εύγλωτα την πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή να υπάρξει συνοχή και σχέση συνεργασία μεταξύ των διαφορών επιπέδων ευθύνη, δημόσια και ιδιωτική. Οι μεταφορέ έχουν και ένα άλλο χαρακτηριστικό που είναι αξιοσημείωτο. Εκεί διασταυρώνονται όλε οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ στην υλοποίησή του. Επιτρέψτε μου να σα αναφέρω κάποιε από τι προκλήσει του μέλλοντο, αλλά από τρει διαφορετικέ οπτικέ γωνίες Πρώτον, λέγοντα ότι οι μεταφορέ βρίσκονται στο κέντρο τη ευρωπαϊκή οικονομική δραστηριότητα, οι μεταφορέ και το σύστημα μεταφορών μα είναι υψηλή ποιότητα και εξασφαλίζουν ανταγωνιστικότητα για την ε, ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία αλλά και ως προς τις θέσεις απασχόλησης ή την ε, οικονομική ανάπτυξη. Οι μεταφορές παίζουν ένα ρόλο ζωτικό και στην αυστηρή τους ε, ε, έννοια και ορισμό, αλλά και γενικότερα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, όπως είπε σωστά η πρόεδρος Ντελή, για το μέλλον του πλανήτη, ε, το πώς θα χειριστούμε τις μεταφορές για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αλλά και όλους τους φορείς που ασχολούνται με την ανάπτυξη του συστημάτων μεταφορών. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με οικονομική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή πρέπει να είναι και βιώσιμη από κοινωνική σκοπιά αλλά και από τη σκοπιά των περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. Οι πολιτικές που υλοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο μέγιστος ε, ε, ο, μάλλον ο πρώτος παράγοντας που καθορίζει τις πολιτικές αυτές και συνυπέγραψε την ε, Συμφωνία των Παρισίων εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Είτε αμέσως ε, χάρη στην Συμφωνία των Παρισίων που θα επηρεάσουν λόγω χάρη μέσω της ΙΑΤΕ την, τις ευρωπαϊκές μια ευρωπαϊκή αρμοδιότητα ή το τι θα γίνει με τον Ευρωπαϊκό ε, Οργανισμό των Θαλάσσιων Μεταφορών, μάλλον με τον Διεθνή Οργανισμό Θαλάσσιων Μεταφορών ε, και τις θαλάσσιες μεταφορές γενικότερα. Οι κλιματικές αλλαγές γίνονται πρώτη μας ε, πρόκληση. Στον τομέα των μεταφορών, νομίζω άλλοι θα τα θίξουν με τρόπο πιο εύστοχο από μένα στη συνέχεια, οι μεταφορές αφορούν και την καθημερινότητα, τη δική σας καθημερινότητα. Οπότε η διάσταση, τέλο πάντων η ευρωπαϊκή δουλειά, θα πρέπει να συσχετιστεί αποτελεσματικά με τη δουλειά που κάνουν οι φορεί και οι αρχέ σε εθνικό επίπεδο για τα θέματα αυτά. Και σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο το ίδιο. Η κυκλοφορία, η μαζική μετακίνηση των πολιτών ε, μέσω σιδηροδρόμων ε, στην, ε, στα αστικά κέντρα, ηλεκτροκίνηση, η καλύτερη χρήση στο μέλλον της ευφυούς ψηφιοποίηση. Όλα αυτά είναι δυσκολίες, οι προκλήσεις, οι στόχοι που χρειάζονται ευρωπαϊκή επεξεργασία. Θα πρέπει λοιπόν και οι πόλεις και οι περιφερειές να αναβλάβουν ευθύνη για την υλοποίησή τους. Οι ίδιοι οι φορείς και οι χρήστες των συστημάτων μεταφορών, εσείς οι ίδιοι δηλαδή. Αυτά και θα ήθελα να ολοκληρώσω παρουσιάζοντας με τρόπο αμεσότερο ενδεχομένω πως η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών λαμβάνει μέρημνα για τους χρήστες και γενικότερα για τους πολίτες με τρία παραδείγματα. Το πρώτο είναι η Ευρωπαϊκή Άδεια, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οδήγησης, με ιδιαίτερα τεχνικές προδιαγραφές και κανόνες, αλλά θα μας επιτρέπει ε, σε όλους να κυκλοφορούμε αποτελεσματικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και ένα τεχνικό εργαλείο για να, γίνει, να λάβει σαν καρκιωστά ε, μια ευρωπαϊκή φιλοδοξία. Η οδική ασφάλεια, που είναι κυρίως εθνική αρμοδιότητα, αλλά με καλύτερες πρακτικές και ευρωπαϊκά εργαλεία, πιστεύω ότι μπορούμε σήμερα να γίνουμε φιλοδοξότεροι και να μειώσουμε τον αριθμό νεκρών, που είναι απαράδεκτος ο αριθμός, στους ευρωπαϊκούς δρόμους και αυτοκινητοδρόμους. Το δεύτερο παράδειγμα είναι οι αερομεταφορές. Η εσωτερική αγορά αερομεταφορών έχει ε, οργανωθεί στη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Εάν σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε με χαμηλό κόστος για περίπου όλους τους πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το επέτρεψε ακριβώς αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι δημιουργήθηκαν και ιδρύθηκαν μια σειρά από αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ενδεχομένως σας επέτρεψαν να είστε εδώ σήμερα το απόγευμα. Αυτή η εσωτερική, η ενιαία αγορά και αυτή αυτή η προσπάθεια να υπάρξει προσφορά στις αερομεταφορέ, ικανοποιητική προσφορά, συνοδεύτηκε και από μεγάλε φιλοδοξίε το δίκαιο περί δικαιωμάτων των επιβατών. Και αυτά χάρη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σα εξασφαλίστηκαν. Νομοθεσία που φυσικά μεταφέρθηκε μετά στην Εθνική Νομοθεσία και εφαρμόζεται από του αερομεταφορεί. Όμω, ελπίζω και το εύχομαι ότι αν ακυρωθούν οι πτήσει σα ή καθυστερήσουν για πολλέ ώρε, θα λάβετε ε, αποζημίωση στην οποία έχετε δικαίωμα ε, και χρηματική πολλέ φορέ για να να αντισταθμιστεί ε, η ζημιά που σας προκλήθηκε και να ισχύσει το δικαίωμα επιβάτου που έχετε. Και θα πω και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσω, ελπίζοντα ότι είμαι μέσα στο δεκάλεπτο, να πω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση των ερχόμενων εβδομάδων, μηνών και ετών είναι να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ ενός τομέα μεταφορών που να είναι αποτελεσματικός, να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και των εταιριών και επιχειρήσεών μας που είναι δραστήριες και σε διεθνές επίπεδο ώστε να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη με περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και προστασία του κλίματος και ταυτόχρονα την πρόκληση της ηλεκτροκίνησης των μεταφορών, κάτι που έχει αναλάβει και το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι, θεσμικοί, όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια σειρά από προτάσει τι ερχόμενε εβδομάδε ώστε να προτείνει εργαλεία για την κινητικότητα με όσο το δυνατόν χαμηλότερες εκπομπές. Ε, σε αυτό το πλαίσιο θα αναθεωρηθούν οι προδιαγραφές για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα, αλλά αυτές οι διατάξεις θα εφαρμοστούν και στα φορτηγά. Φορτηγά που αυτή τη στιγμή ε, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς, ως προς τα πρότυπά μας. Θα ενισχυθούν οι, υποδο, οι επενδύσεις στις υποδομές για να μπορέσουν οι ηλεκτρικές ε, μεταφορές να επεκταθούν στην Ευρώπη, στα αστικά κέντρα αλλά και στους μεγάλους άξονες μεταφορών τους διακρατικούς άξονες και θα κοιτάξουμε να διευκολύνουμε την δημιουργία των ε, ε, σταθμών ηλεκτρικής επαναφόρτησης. Αυτές είναι φιλοδοξίες οι οποίες θα πρέπει σαφώς να συνοδεύονται από την προσπάθεια καινοτομία της αυτοκινητοβιομηχανίας μας που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο καλούν να αξιοποιήσουν αυτή τη φιλοδοξία για να δημιουργήσουν μια βιομηχανική παραγωγή ελπιδοφόρα σεβόμενη τι κοινωνικέ και περιβαλλοντικέ προκλήσει. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα πρώτα λόγια. Να μερικέ πρώτε ιδέε για να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο τη συζήτηση. Αλλά πριν ανοίξει αυτή η συζήτηση, να πω ότι η Επιτροπή στην οποία εργαζόμαστε έχει και εγώ ίδια έχω στην διάθεσή μου μία γραμματεία. Η γραμματεία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί που με συνδράμουν, βρίσκονται στο πλευρό μου η Σουζάν, ε, το επίθετό της μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, έτσι την αποκαλώ εγώ, είναι επικεφαλής ε, της υπηρεσίας, τμήματάρχης, με κοιτάει με κοκκινισμένη και σκέφτεται πω τι θα πει τώρα. Είναι λιγάκι αυτοί που μας λύνουν τα χέρια οι άνθρωποι αυτοί Ποτέ δεν μπορεί κανείς να τους ευχαριστήσει αρκετά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που χάρη σε εσά τσουλάει αυτή η Επιτροπή. Διότι είναι πολλά τα κείμενα που περνάνε από τα χέρια σας και βρισκόμαστε σε μια Επιτροπή όπου πραγματικά το 100% των ε, εκθέσεων που περνάνε από εμά είναι νομοθετικού χαρακτήρα. Έχουν άμεσο αντικτύπο στη ζωή σας δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ τη Γραμματεία. Έχουμε και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι πάντα παρόντες και εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Τι είναι το Συμβούλιο, ε, είναι η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη. Είναι πάντα παρόντος. Όχι, στην προηγουμένη περίπτωση δεν είναι. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συζήτηση και έχετε το λόγο για να μας πείτε ποιες είναι οι προσδοκίες σας, ποια είναι τα θέματα που θα θέλατε να θίξουμε. Βέβαια, το πιο δύσκολο είναι να λάβει το λόγο ο πρώτος. Έχετε το λόγο. Πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο που είναι μπροστά σας Καλημέρα σε όλους και όλες. Ε, πράγματι δεν είναι εύκολο να είναι κανείς ο πρώτος ομιλητής εδώ και 15 χρόνια στη Γαλλία ε, ζούμε την απορρίθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών, πρώτο και δεύτερο πακέτο για την μεταφορά των εμπορευμάτων και θα ήθελα να μου πείτε ποιες, ποιος είναι ο απολογισμός του συσχετισμού οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών μέσα στα πλαίσια του πρώτου και δευτέρου πακέτου. Το όνομά σας παρακαλώ. Ολιβιέ λέγομαι. Θα θέλαμε λοιπόν έναν απολογισμό αυτού, αυτής της απορρίθμισης ε, του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων. Γιατί είχαμε να κάνουμε προηγούμενα με ιστορικούς φορείς και βλέπουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν άκρατο φιλελευθερισμό. Ως προς τις καθημερινές μεταφορές στις χώρες που ε, ε, γνωρίζουν μία γεωγραφική απόκληση, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα το περιβάλλον. Ζούμε σε πόλεις που χτίστηκαν το 19ο αιώνα, όπου δεν υπήρχε θέση για τα αυτοκίνητα βλέπουμε ότι έχουν γίνει μελέτες και από το 2000 και μετά η χρήση των, των οχημάτων έχει αυξηθεί καθώς και το πλάτος τους κατά 14 εκατοστά. Υπάρχει κάποια νομοθεσία, ευρωπαϊκή νομοθεσία για το μέγεθος των οχημάτων, γιατί στις ευρωπαϊκές πόλεις δεν μπορούμε να παρκάρουμε πλέον. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις, ε, χώρες, για τις πόλεις της Βόρειας Γαλλίας ή το Βέλγιο. Ευχαριστούμε, Ολίβιε. Τέταρτο πακέτο, σιδηροδρομικό πακέτο, λοιπόν, ε, οδηγεί σε απελευθέρωση ή όχι ως προς τις καθημερινές ε, μεταφορές και τα, ε, τις κλιματικές αλλαγές. Τις λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά και μιλήσατε και για τα οχήματα και το μέγεθός τους. Τέσσερις είναι οι ερωτήσεις σας. Ε, άλλες ερωτήσεις από άλλους ομιλητές έχετε το λόγο. Να μας πείτε καταρχήν ποιος είστε, από πού έρχεστε. Ε, είμαι μηχανικός και έρχομαι από τη Ρουμανία. Μπορείτε. Ε, έρχομαι από τη Ρουμανία, όπως είπα, και είμαι καθηγητής, μηχανικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Οπωσδήποτε οι μεταφορές είναι ύψης της σημασίας και θα είχα κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Δυστυχώς τα οδικά δίκτυα, το δικό μας οδικό δίκτυο δεν είναι ανεπτυγμένο στη Ρουμανία. Και γι' αυτό γνωρίζουμε και μεγάλο αριθμό ατυχημάτων και γι' αυτό θα έπρεπε να προβούμε σε μια πιο ε, οικολογική χρήση των μεταφορών, δηλαδή όσο αφορά τα εμπορεύματα θα έπρεπε να μεταφέρονται με, από τους σιδηρόδρομους και να μην μεταφέρονται οδικώς. Θα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε και εναλλακτικέ πηγές ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα Επίσης δεν υπάρχει μία σωστή ε, ε, ρύθμιση του πλαισίου της ενέργειας και των μεταφορών για να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, διότι υπάρχουν ε, χώρες όπου η έμεση φόρη είναι πολύ υψηλή στα καύσιμα, κάτι το οποίο οδηγεί σε αθέμητο ανταγωνισμό. Θα περιοριστώ σε αυτές τις τέσσερις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένας, ακόμα ένας ομιλητής για αυτό το γύρο. Καλημέρα. Μπορείς Βενσάν, είμαι εδώ ως πολίτης και έχω ξεκινήσει μια startup στον τομέα της ποδηλασίας ε, bike.fr που ε, σχετίζεται με την κοινή χρήση ποδηλάτων από ιδιώτες. Μιλάμε λοιπόν για ένα τομέα καινοτομία στις μεταφορές και θα πρέπει να δούμε πώς ε, η καινοτομία εφαρμόζεται έμπρακτα, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για μικροϋποδομές όπου υπάρχει πολύ ταλέντο αλλά περιορισμένα μέσα και εξού και ο πολυσχηδής χαρακτήρας των ε, μεταφορών. Έχουμε να κάνουμε με περιορισμένες υποδομές και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολλούς εμπειρογνώμονες για να χειριστούν τα θέματά μας. Θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές αλλά και αποτελεσματικοί στον τομέα της ε, καινοτομίας έτσι ώστε ε, να γίνονται σωστές ε, χρηματοδοτήσεις και να φτάνουμε στον απότερο στόχο ως προς την καινοτομία, έμπρακτη καινοτομία και προς τα πάνω. Καινοτομία προς τα πάνω, ναι. Τι θα κάνουμε έτσι ώστε οι νεοσύστατες εταιρείες, οι startups να έχουν ε, πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτή στην ουσία είναι η ερώτησή σας. Εμείς έχουμε κάνει ένα κύκλο διαπραγματεύσεων με επιχειρήσεις στην Αλσατία, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, περιορισμένες δυνατότητες, ιδιαίτερα προς την επιχείρηση BEA σε σχέση με τη χρήση των ποδηλάτων. Και αυτό είναι και ένα πολιτικό ερώτημα. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει παγκοσμιοποίηση σε αυτό το θέμα ως προς τους ε, φορείς πρόθεσης. Έχουμε εγκεφάλους, ταλέντα, και υποδομές. Θα πρέπει όμως όλα αυτά να τα συντονίσουμε γιατί υπάρχει μία δυσλειτουργία σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πραγματιστές. Ωραία. Θα αρχίσουμε να απαντάμε σε ερωτήσεις σας. Να τις επαναλάβω. La question du ως προς το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο υπάρχει πραγματική ε, απελευθέρωση καθημερινές μεταφορές. Λαμβάνουμε υπόψη στην Επιτροπή μας τις καθημερινές μεταφορές και το περιβάλλον, η θέση των οχημάτων. Ποια είναι η θέση των οχημάτων, ιδιαίτερα ως προς το μέγεθός τους. Και στη συνέχεια δεν θα πρέπει να ε, μιλήσουμε για τη μεταφορά εμπορευμάτων, πρέπει να γίνεται σιδηροδρομικός και όχι οδικός. Ως προς την ε, ανταγωνιστικότητα και τους φόρους καυσίμων, πώς νομοθετούμε. Καθώς ε, και όσο αφορά την καινοτομία, πώς την αντιμετωπίζουμε και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποιος θα ήθελε να ε, αρχίσει να απαντά. Ο κύριος Βίμ Βαντερκάμπ και μετά ο κύριος Τελίτσκα. Έχετε το λόγο. Θα μιλήσω Ολλανδικά, ε. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο. Έχουμε τέσσερα πακέτα. Αυτό εγκρίθηκε πρόσφατα, αλλά πρέπει, για να είμαστε ειλικρινεί, να πούμε ότι τα καράτη-μέλη ακόμα τρενάρουν, θα έλεγα, την εφαρμογή. Και συγκεκριμένα η SNCF, ε, η γαλλική κρατική σιδηροδρομική εταιρεία, πρέπει να εφαρμόσει το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο και από ό,τι φαίνεται θα αργήσει, δεν είναι υπέρ του ανοίγματο της αγοράς. Λοιπόν, εδώ πέρα κάνουμε δύο είδη νομοθεσίες. Οδηγίες και κανονισμούς. Αλλά οι οδηγίες πρέπει μετά στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στην Χάγη, να μεταφερθούν σε εθνική νομοθεσία και κάπου εκεί πέρα κάτι χάνεται από το ευρωπαϊκό ιδέο. Και έρχομαι άρα στην αρχή της επικουρικότητας γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε ποτέ για συγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ σε πόλεις και χωριά. Αυτό είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Γιατί καμιά φορά δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, είτε μιλάμε για startups είτε για οτιδήποτε άλλο. Έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πρόγραμμα για startups, για νεοφυείς επιχειρήσεις, ειδικά στον τομέα της πληροφορικής, οπότε θα έλεγα κάντε ερωτήσεις ελεύθερα και αιτήσει βεβαίως. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ριβόνταλόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση για αυτό το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, το οποίο όντω ψηφίστηκε στην Επιτροπή Μεταφορών και από το Ευρωκοινοβούλιο. Όμω το Ευρωκοινοβούλιο είναι πολιτικό θεσμικό όργανο. Οι πολιτικέ ομάδε εκφράζουν την άποψή του και να υπενθυμίσω ότι οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε δεν είχαν υπερψηφίσει την ε, απελευθέρωση των δημόσιων υπηρεσιών, διότι ως προς την απελευθέρωση του σιδηροδρομικού δικτύου χρειαζόμαστε κοινωνικές εγγύησεις, κοινωνικά εχέγγυα που ε, δεν προβλέπονται στις υποχρεώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και τη διατήρηση γραμμών όταν δεν είναι αναγκαστικά οικονομικός κερδοφόρες. Αυτό ήταν σημαντικό για μας, διότι το θέμα της κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης για μας ήταν πολύ σημαντικό. Ως προς το θέμα μεταφορές και περιβάλλον, αυτό είναι ένα άκρο πολιτικό ζήτημα που απασχολεί την Επιτροπή μα, την Επιτροπή Μεταφορών. Το συζητήσαμε μόλι σήμερα το πρωί. Βλέπουμε εκεί ότι οι στόχοι, οι φιλόδοξοι στόχοι των συμφωνιών των Παρισίων τη COP21 ε, δεν είναι πάντοτε ε, γραμμή που ακολουθούν όλε οι ομάδε. Και εκεί όμω αγωνιζόμαστε ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, να μπορέσουμε να μειώσουμε το 30% που είναι η ρήπανση, η ρήπανση που προκαλείται από τι μεταφορέ. Πρόκειται για ένα challenge, μια πρόκληση πολύ σημαντική. Ε, εκεί πρέπει να υπάρξουν βελτιώσει, αλλά πρέπει να πάμε και μακρύτερα στις προτάσεις μας, την νομοθεσία που προτείνουμε δηλαδή, και να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να σέβονται αυτήν την ε, γραμμή την στάση συμπεριφορά που οι ίδιοι ενέκριναν στην διάσκεψη των μερών 21, την Συμφωνία των Παρισίων. Πρόκειται λοιπόν για μια άκρο πολιτική συζήτηση, όπου στο Κοινοβούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζεται μέσω των διαφορετικών πολιτικών ομάδων το βάρο του στι ψηφοφορίε. Έγινε το 2014, θα γίνει και το 2019. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τι εκλογέ, ώστε ο πολιτικό προσανατολισμό που ακολουθεί η Ένωση να ανταποκρίνεται στι προσδοκίε σα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κυρία Ριβονταλόν, ο κύριο Τελίντσκα. Uh, Θέλουμε να έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση, αλλά θα είμαι πολύ σύντομο ε, σύντομος ως προς την απελευθέρωση του πακέτου σιδηροδρόμων. Ο κύριος Βαντερκάμπ είπε ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν τα καταφέρνουν αρκετά καλά ως προς την εφαρμογή του πακέτου. Χρειαζόμαστε καλύτερη εφαρμογή. Θέλουμε την απελευθέρωση, θέλουμε να έχουμε μια λειτουργική εσωτερική αγορά, δεν θέλουμε να είμαστε επιλεκτικοί και μας, ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν τα ωφέλη, η ανάπτυξη και επιλογές του καταναλωτή. Εγώ είτε ως ε, άτομο είτε ως ε, επιχείρηση θέλω να διαθέτω την ε, δυνατότητα επιλογής και θα πρέπει να άρουμε όλες τις στενοπούς της απελευθέρωσης. Διαφωνώ με τους σοσιαλιστές γιατί θεωρώ ότι οι προτάσεις των σοσιαλιστών δεν είναι οι καλύτερες δυνατές ως προς τη, τα οχήματα και το μέγεθός τους. Θέλουμε να, να ρυθμίσουμε αυτό το πλαίσιο, μα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Διαφορετικά θα πρέπει να ρυθμίσουμε τα πάντα, το μέγεθος που έχουν οι ρόδες, τα καθίσματα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή εκεί όπου υπάρχει προστιθέμενη αξία. Υπάρχουν θέματα που αφορούν την εσωτερική αγορά, το περιβάλλον, καθώς ε, και το κοινωνικό κεκτημένο ως προς τους έμεσους φόρους στα καύσιμα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού η φορολόγηση ως προς την φορολόγηση και τους έμεσους φόρους, τα κράτη δεν θέλουν να προβούν σε εναρμόνιση πάντα. Ως προς τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της καινοτομίας, ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, να είμαστε πιο φιλικοί προς το χρήστη, αυτό αφορά την Κομισιόν αλλά ναι. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει όμως επιτελεστεί πρόοδος και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Ε, δεν υπάρχει απάτη ή απορρίθμιση, αλλά πολλές φορές ο διοικητικός φόρτος αφορά το εθνικό επίπεδο. Δηλαδή σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζουμε τα, όλα αυτά τα θέματα αλλά με μεγαλύτερη περιπλοκότητα. Λοιπόν, θα βάλουμε το χρονόμετρο, διαφορετικά ο καθένας θα μιλάει τρία λεπτά και θα πρέπει οι πολίτες να έχουν το λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την απελευθέρωση. Θεωρώ επί της αρχής ότι βλέπουμε παραδείγματος χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο που η απελευθέρωση έχει αρνητικές συνέπειες για τους σιδηρόδρομους που ο ανταγωνισμός ή μάλλον η ανταγωνιστικότητα χάθηκε και σε άλλες χώρες βλέπουμε υπερβολικό προστατευτισμό που οι σιδηροδρομοί έχασαν την ανταγωνιστικότητά τους ε, ειδικά στα διασυνοριακά δρομολόγια. Οπότε ε, ακούστηκε ότι χρειάζεται μια υψηλότερη τιμή κλίματος. Ε, πρέπει δηλαδή να γίνει φτηνότερο να ταξιδεύει κανείς με το τρένο και ακριβότερο να παίρνει κανείς αεροπλάνο ή το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Βεβαίω καλό θα ήταν να έχουμε ε, μεταφορές εμπορευμάτων με το τρένο. Έχουμε 100% 100 των σιδηροδρόμων πληρώνει τέλη στην Ευρώπη ενώ 1% των δρόμων του οδικού δικτύου στην Ευρώπη έχει διόδια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, απελευθέρωση εγώ είμαι κατά των μονοπωλίων, κρατικών ή ιδιωτικών. Έπρεπε να κλείσουν ε, τη γραμμή μεταξύ Κάρστ ε, και Σβέλφατ, ε, γιατί είχαν μόνο 500 επιβάτες τον χρόνο. Και τελικά, όταν ξαναξεκίνησε, έχουν 32.000 επιβάτες αν επικρατούσε τελικά η Deutsche Bahn, αυτές οι 32.000 θα έπαιρναν το αυτοκίνητο. Σας ευχαριστώ. Κύριος Κίλωνεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κάποιες απαντήσεις που ίσως να μην έχουν ακόμα δοθεί. Καλό ερώτημα για αυτές τις startups είναι ακριβώς ε, το θέμα των startups και τα λοιπά δεν είναι εύκολο γιατί το lobbying πάντα εκπροσωπεί τι μεγάλες ε, εταιρείε ε, και είναι δύσκολο να δούμε πώς θα βοηθήσουμε αυτούς που τώρα ξεκινάνε την επιχείρησή τους και πώς μπορούμε να κάνουμε, να επιφέρουμε αλλαγές στις πόλεις, πώς θα χρησιμοποιήσουμε λιγότερα αυτοκίνητα. Χρειαζόμαστε μεγάλες αλλαγές πρώτα απ' όλα μεταξύ των αυτιών, κάπου στον εγκέφαλο δηλαδή. Δηλαδή χρειάζομαι αμάξι, μήπως μπορώ να το μοιραστώ. Μπορεί να περάσουμε στην κινητικότητα ως υπηρεσία. Και μετά όταν βρούμε τις βέλτιστες πρακτικές στην πόλη, πώς μπορούμε να τις διαμοιράσουμε και να δοθεί η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συστήματα χαμηλών εκπομπών και τέτοια πράγματα. Σαν μέσα μαζικής μεταφοράς, ε, την, την οικονομία του διαμοιρασμού και δεν μπορούσα να λέω κι άλλα, αλλά έχει τελειώσει ο χρόνος μου. Σας ευχαριστώ κύριε Κίλονεν. Ερωτήσεις από το Twitter. Madame la Présidente, alors il y a une grande activité sur Twitter. Ε, Υπάρχει πολλή δράση στο Twitter. Λάβαμε ερωτήσει για πολλά θέματα, αλλά κυρίω το αυτόνομο όχημα έχει λάβει πολύ. Ε, πολλές ερωτήσεις. Ο κύριος Μενιέ, δικηγορός, μας λέει πώς η Ευρώπη θα αναδείξει τους επόμενους πρωταθλητές των αυτόνομων οχηματών ο κύριος Μπρεβεσάλ λέει τι θα γίνει με τις startup επιχειρήσεις που μας ρωτούν πώς θα μπορέσουν τα αυτόνομα οχήματα να γίνουν ε, γιοταχή. Επίσης, ε, κάποιος από το νόμιλο Airbus μας λέει πώς θα ε, συνδυάσουμε το αυτόνομο όχημα με την ε, μοιρασμένη οδήγηση και πώς θα αποφύγουμε τις επιθέσεις σε περιορισμένα κοινωνικά πλαίσια. Όλα αυτά σε σχέση με το αυτόνομο όχημα και κάτι άλλο από τον Ματιέ από τι αστυνομικέ δυνάμει που μας λέει σε περίπτωση ατυχήματος ένα αυτόνομο όχημα θα πρέπει να επιλέξει θυσία μεταξύ της ζωής του ε, οδηγού ή του πεζού σε περίπτωση που ο πεζό του προκαλεί. Ευχαριστώ. Ερωτήσει από το Twitter. Θα ακούσω άλλη μια ερώτηση από την κυρία εκεί, μάλλον από τον κύριο που σήκω στο χέρι. Παρακαλώ. από τη Γερμανία. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Η νομοθεσία έγκρισης τύπου λέει πως ε, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση και του software και αν αλλάξει το software θα πρέπει να υπάρξει ξανά έγκριση τύπου. Δεν ξέρω εάν ε, γνωρίζετε αν ε, μπορεί να αλλάξει κάτι τέτοιο στο μέλλον και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί αυτό στο μέλλον δεδομένων και των αναβαθμίσεων που γίνονται στο software ε, για να μπορούν και οι οργανισμοί τεχνικού ελέγχου να πιστοποιούν ότι πράγματι το αυτοκίνητο κάνει αυτά τα οποία πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σε σχέση με τα αυτόνομα οχήματα, τους κινδύνους και τα ατυχήματα, πιστοποίηση επίσης των ε, οχημάτων και πώς θα έχουμε κολοσσούς startups στην Ευρώπη και πώς θα μπορέσουμε να τους παρακολουθήσουμε. Πολίτες, προσπαθούμε να προτρέξουμε του μέλλοντος. Γι' αυτό η Επιτροπή μας δημιούργησε Ευρωπαϊκό Βραβείο για startups της κινητικότητας. Δεν θα πρόκειται για ένα δίπλωμα ή ένα ευρωπαϊκό κύπελο. Απλώς θα θέλαμε να προωθήσουμε τις νεοσύστατες ε, εταιρείε. Ξέρετε το BlaBlaCar. Αύριο θα έχουμε και άλλους κολοσσούς, γι' αυτό κατά τα τέλη του Νοεμβρίου όλες οι startups της, στο τομέα της κινητικότητας θα πρέπει να υποβάλουν τα σχέδιά τους. Θα έχουμε μία εξεταστική επιτροπή επτά από 7 μέλη. Ε, θα λάβουμε υπόψη μία startup από το Βερολίνο, την Υπουργό της Εστονίας υπεύθυνη για την ψηφιοποίηση και στις 22 θα έχουμε αυτό το έπαθλο, δηλαδή θα επιλέξουμε 10 νεοσύστατες εταιρείες που ασχολούνται με θέματα κινητικότητας. Δηλαδή δεν μιλάμε παρά για μία ενιαία κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς που περιλαμβάνει τους πάντες. Επίσης έχουμε και το κριτήριο της χρηστικότητας και της χρησιμότητας της κινητικότητας. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την οδική ασφάλεια. 126.000 θάνατοι στα οδικά μας δίκτυα εδώ στην Ευρώπη και χιλιάδες τραυματίες. Δεν το δεχόμαστε πλέον αυτό. Γι' αυτό θα δημιουργήσουμε αυτό το βραβείο για να έχουμε νέους κολοσσούς startups που ασχολούνται με την ψηφιοποίηση στον τομέα της κινητικότητας. Γιατί τι γίνεται όταν ανακύπτουν τότε αποχωρούν στη ΣΥΠΑ, προς τη ΣΥΠΑ και δεν παραμένουν στην Ευρώπη. Εμείς θα θέλαμε να παραμείνουν στην Ευρώπη και θέλουμε να τις παρακολουθήσουμε ως προς τα αυτόνομα οχήματα. Κύριε Ερτούγκ, Μπορείτε να μας πείτε σε περίπτωση ατυχήματος ποιος είναι ο υπεύθυνο. Ε, ε, είναι το λογισμικό, ο οδηγός, η αυτοκινητοβιομηχανία. Τι κάνουν και οι ασφάλειες σε αυτή την περίπτωση. Αυτά τα θέματα μας απασχολούν εδώ και στην, ως προς την πιστοποίηση των ε, οχημάτων και η κυρία Ρεβόντα Λόν θα μας απαντήσει παράλληλα γι' αυτό το σε αυτό το ερώτημα. Ο κύριο Ερτούγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση πρώτα απ' όλα για το δικτύωμένο και αυτόματο αυτοκίνητο. Πρέπει να γίνει μια διάκριση εδώ πέρα μεταξύ των διαφόρων φάσεων εξέλιξης που έχουμε μεταξύ ημιαυτόματων και αυτομάτων αυτοκίνητων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο επίπεδο 2 έχουμε ήδη συστήματα που βοηθούν τον οδηγό ε, με τα οποία α, μπορούμε να οδηγήσουμε. Είτε μιλάμε για στήματα αυτόματου, φρεναρίσματος ή αυτά που κρατάνε το αυτοκίνητο στη λωρίδα είναι κάποιο είδους αυτόνομη οδήγηση. Αυτό το οποίο εννοούν οι πολίτες είναι το μελλοντικό όραμα ότι κάθεται κανείς στο αμάξι και αυτό μας πηγαίνει μόνο του. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα αλλά είμαστε πάρα πολύ κοντά όσον αφορά το επίπεδο 3. Δηλαδή να παίρνουμε τα χέρια από το τιμόνι όταν είμαστε στον αυτοκινητόδρομο, στο μποτιλιάρισμα. Οπότε ξέρει το αυτοκίνητο πότε πρέπει να ξεκινήσει και να σταματήσει. Υπάρχουν πράγματα βέβαια που πρέπει να ξεκαθαρίσουν και ρυθμιστικά νομικά ζητήματα, δηλαδή που αφορούν την αστική ευθύνη, τις υποδομές, ε, την κοινωνική αποδοχή. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Γι' αυτό ελπίζω η Κομισιόν ως εκτελεστικό προσεχώς ε, να μας κάνει μια πρόταση για το πώς μπορούν να ρυθμιστούν αυτά τα πράγματα και πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ερευνούν ε, το θέμα και βεβαίως χρειαζόμαστε μια άλλη διαδικασία έγκρισης τύπου, χρειαζόμαστε και νέες δυνατότητες για το πώς ε, θα γίνουν οι έρευνες, τι θα γίνει με τις άδειες, όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν. Αλλά μπορώ να σας πω ότι η αυτόνομη και δικτυωμένη οδήγηση είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία αφενός για να γίνει πιο ευχάριστη η κινητικότητα αλλά και για να μειωθούν ξεκάθαρα τα α, Ευτό Γι' αυτό εγώ είμαι μεγάλος υπέρμαχος ε, της αυτόνομης και δικτυωμένης οδήγησης. Ευχαριστούμε, αλλά δεν μας είπατε με τι θα τρέχει το αυτόνομο όχημα αύριο. Με τι θα κινείται. Α, τώρα άμα ανοίξουμε αυτό το βαρέλι όπως λέμε στη Βαβαρία λοιπόν είναι μια ακαθόδης ε, πολιτική απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί Δεδομένου και του σκανδάλου με το ντίζελ, από ό,τι φαίνεται, θα τεθεί το ερώτημα του αν θα διατηρηθεί η τεχνολογία ντίζελ ή γενικά οι κινητήρες σε εσωτερικές αν θα πάμε σε ηλεκτρικούς κινητήρες ε, ή σε κινητήρες υδρογόνου ή σε κάποια άλλη τεχνολογία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή, αν είναι π.χ. ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα που θα φορτίζουν, πόσες ε, θέσεις εργασίας ε, υπάρχουν σήμερα στην ε, βιομηχανία, πόσα από αυτές θα χαθούν. Μιλάμε για 7 θέσεις εργασίας πάνω σε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης που θα αντικατασταθούν από μία θέση εργασίας σε ηλεκτρικό κινητήρα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια μεταβατική φάση για να γίνει αυτή η μετάβαση. Και όπως σας είπα αυτό το θέμα δεν ε, μπορεί ακόμα να απαντηθεί οριστικά, θα απαντηθεί στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κύριε Ερτού. Ευχαριστούμε κύριε Ριβονταλόν. Θέλετε να πείτε και εσεί κάτι. Ναι, ένα λεπτό μόνο. Για το θέμα τη πιστοποίηση. υπάρχει ένα νομοθετικό κείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή συζητιέται σε επίπεδο τριμερού διαλόγου μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπή και Συμβουλίου δηλαδή για τι νέε προτάσει σχετικά με την ενίσχυση τη διαφάνεια των ελέγχων και των κυρώσεων σε περίπτωση μη και επιτέλου, αυτή τη στιγμή αρχίζουν ε, τα τεστ σε συνθήκε πραγματική οδήγηση που θα μα επιτρέψουν να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Οι εθνικές ε, πιστοποίησης θα παίξουν εδώ καθοριστικό ρόλο, όμως σε κάθε περίπτωση διατηρούμε και αυτό ήταν μέρος των προτάσεων που είχαμε κάνει στα, στο επίπεδο της, της Εξεταστικής Επιτροπής για τον Dieselgate, διατηρούμε τις προτάσεις για, ε, μια, για έναν εξάρτητο ευρωπαϊκό οργανισμό για να παρακολουθεί και να ε, οργανώνει κεντρικά τι διάφορε εθνικέ αρχέ που είναι υπεύθυνε για την εξουσιοδότηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τελίντσκα. Ευχαριστώ. Μπορώ να απαντήσω δύο ερωτήσεις ε, με, με περίπου πάνω κάτω μια απάντηση για το πώς θα βρούμε τους πρωταθλητές του αύριο. και να βεβαιωθούμε ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα θα είναι μια πραγματικότητα και τι είδου καύσιμα θα καταναλώνουν. Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζεται να πάρουμε εμεί την απόφαση για τον καταναλωτή. Δεν είναι αυτό ο ρόλο μα. Ο ρόλο μα είναι να μην ευνοήσουμε κανένα στην αγορά περισσότερο από άλλον. Κάποιον που δεν θα συμμορφώνονται μάλιστα με κανόνε και προδιαγραφέ που εμεί αποφασίσαμε. Αυτό είναι κάτι που η αγορά, βάσει του ρυθμιστικού περιβάλλοντο που θα δημιουργήσουμε, θα το λύσει τη Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη πρέπει να βεβαιωθούμε, όπω είπε και ο πρόεδρος, ότι οι ταλαντούχοι άνθρωποι δεν θα ξεκινήσουν να πάρουν τα μπογαλάκια τους να πάνε στο Silicon Valley, αλλά θα μείνουν εδώ, εδώ να προσφέρουν το ταλέντο τους. Αυτή είναι η θετική πρόκληση. Πρέπει να μείνουν να φτιάξουν startup Θέλουμε εμεί βέβαια να προλυάνουμε το έδαφο, να είναι γόνιμο για τη startup, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν, να μεγαλώσουν και να γίνουν πρωταθλήτριε. Δεν είναι θέμα μεγέθου, είναι θέμα του πόσο συμβατό θα είναι το ρυθμιστικό περιβάλλον που θα φτιάξουμε. Το ίδιο είναι και αυτό που ισχύει για τα αυτοκίνητα. Είτε είναι ηλεκτροκίνητα, είτε υδρογονοκίνητα, είτε ολική ενέργεια, είτε με πανιά. σω κάποτε στο μέλλον. Δεν ξέρουμε πώ θα γίνει. Δεν είναι δική μα η απόφαση όμω. Είναι κάτι που η αγορά, ο ανταγωνισμό και η ζήτηση θα το κάνουν. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Τελίντσκα ο κύριος Πακέτ πρέπει να φύγει. Θα σας δώσω δύο λεπτά. Προσπαθήστε κι εσείς να απαντήσετε κάπως εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύνολο των ερωτήσεων που ήταν κάτι παραπάνω από εύστοχες. Ευχαριστώ. Θα επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα. Καταρχήν, μεταφορά των εμπορευμάτων σιδηροδρομικός και φυσικά το τέταρτο πακέτο καλύπτει τη διαλειτουργικότητα και δημιουργεί τους όρους έτσι ώστε τα εμπορεύματα να μεταφέρονται με κατά ανταγωνιστικό τρόπο και φυσικά θα υπάρχουν και διάδρομοι για το μέλλον των μεταφορών των εμπορευμάτων όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές τους. Θέλουμε λοιπόν τα εμπορεύματα να μεταφέρονται με, μέσω σιδηροδρόμων παρά να χρησιμοποιούνται τα οδικά δίκτυα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσαρμοστούν σε σχέση με την ε, καινοτομία και τα startups. Με ε, έχει εκπλήξει ευχάριστα το βραβείο σας το βραβείο που ορίστηκε τώρα και φυσικά αυτό που έχει σημασία είναι το κατά πόσο οι νεοσύστατες αυτές εταιρείες κάνουν ένα scaling up. Ως προς την χρηματοδότηση, η Κομισιόν προβλέπει άμεσες χρηματοδοτήσεις που βέβαια ε, δεν καλύπτουν πάντα τις ανάγκες των ε, startups και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προωθούμε την ε, έρευνα μέσα στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 έτσι ώστε να αυξήσουμε την χρηματοδότηση για να περάσουμε από τις startups στις ε, επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε σχέση με το αυτοματοποιημένο όχημα φυσικά υπάρχουν ε, πολλές ε, ενδυνάμει δυνατότητες εργαζόμαστε επί του θέματος και στην Κομισιόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ρυθμίσουμε τον τομέα αυτό γιατί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αλλά θα προωθήσουμε ένα ε, πλαίσιο λειτουργίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πακέ. Θα σας δώσω και πάλι το λόγο. Ο κύριος το βάθος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, Νταβίτ Προυβέ από την ε, ΣΕΖΕΤΕ ε, θα ήθελα να παρέμβω στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Σήμερα όλοι οι τομείς μεταφοράς πλήττονται από το κοινωνικό ντάμπινγκ και βλέπουμε ότι στις δημόσιες μεταφορές η, κατάσταση είναι τραγική. Γίνεται ένας αγώνας ντάμπινγκ σε σχέση με την ασφάλεια, τα προσόντα, και έλλειψη ανθρωπίνων πόρων και υπάρχει έλλειψη ανθρωπίνων πόρων γιατί όπως είπατε δεν μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιεί μία εφαρμογή στο κινητό του. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ε, προωθούν το κοινωνικό dumping καθώς και το φορολογικό dumping. Προβάλλεται επίσης dumping και στον τομέα της ασφάλειας. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε μια πολύ ωραία νομοθεσία, αλλά θεωρώ ότι και οι δύο πλευρές φέρνουν μεγάλη ευθύνη, και η ευρωπαϊκή και η κρατική. Ως προς τα περιβαλλοντικά, αν δεν θέλουμε να υπάρχει ρήπανση, θα πρέπει να αναλάβουμε το κόστος και να μην προβαίνουμε σε εξωτερικές αναθέσεις, διότι οι οδικές και οι σιδηροδρομικές μεταφορές καταβάλουν το κοινωνικό τίμημα. Και αυτό το βλέπουμε και έναντι των χρηστών. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλος. Σούβατ από την Γερμανία. Έχω δύο ερωτήσεις. Έχω δύο ερωτήσει. Λοιπόν, η πρώτη αφορά την αυτόνομη οδήγηση. Ποιε είναι οι προθέσει και ποια είναι η κατάσταση των νομικών προσαρμογών της ε, Σύμβασης της ε, Βιέννης ε, που υπάρχει από το έτος 1968 και δεύτερον θα υπάρξουν νέες δυνατότητες για την επικοινωνία ανθρώπου και τεχνολογίες οι οποίες περιορίζονται αυτή τη στιγμή από τις νομικές διατάξεις. Τι προθέσεις έχετε ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο μεγάλες ερωτήσεις το θέμα του κοινωνικού dumping και δική σας. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους να πω ότι όλοι σε αυτή την Επιτροπή συμφωνούμε ότι το κοινωνικό dumping είναι αυτό που δηλητηριάζει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όλοι επ' αυτού συμφωνούμε. Απλώς μετά έχουμε διαφορετικούς προσανατολισμούς πώς θα ε, ορίσουμε και τι κανόνες θα εφαρμόσουμε κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ. Το πραγματικό ερώτημα είναι σήμερα θα προωθήσουμε την νομοθεσία προς την κοινωνική Ευρώπη με μεγάλους κανόνες, ε, με ελάχιστο μισθό, με ειδικέ προδιαγραφές για την ασφάλεια των εργαζομένων. Άνωθεν είμαστε ικανοί να το κάνουμε αυτό. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Απέναντί μας όμως έχουμε το Συμβούλιο, την ομάδα των αρχηγών και των κυβερνήσεων που δεν έχουν αναγκαστικά τι δικέ μα απόψεις και πολλέ φορέ μπορεί να επικροτήσουν. Ω προ το κοινωνικό λοιπόν dumping, εργαζόμαστε επί. και με συγχωρείτε που θα γίνω λίγο τεχνοκράτησα εδώ, αλλά δεν επιλέγω εγώ του όρου. Εδώ εργαζόμαστε με πακέτα ε, δέσμη Έχουμε το πακέτο για τα σιδηροδρομικά, το πακέτο για την κοινοτικότητα, όπου το κοινωνικό ντάμπινγκ είναι από τι μεγαλύτερε προκλήσει. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ναι, να φροντίσουμε αύριο να αγαπάει ο κόσμο πάλι το τρένο. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει σήμερα κανεί μια low cost, low cost, ακόμη και αν κάποιε εταιρείε δεν σέβονται καθόλου του κανόνε, δεν θα πω ποιε, δεν θα τι κατονομάσω, αντί να πάρει κανείς το τρένο. Και ωστόσο το τρένο είναι ε, εποφελές για όλους. Και για τον επιβάτη και για το κλίμα. Και για την απασχόληση. Άρα πρέπει να δώσουμε έμφαση και στο τρένο. Το θέμα της ανταγωνιστικότητας και του ανταγωνισμού. Της του φορολογικού ανταγωνισμού, έξωθεν κυρίως, δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Κάποιοι τομείς είναι πιο ε, ακριβή από άλλους. Δεν είναι λογικό οι μεταφορέ μεταφορές να μην φορολογούνται λίγο παραπάνω από άλλους τομείς. Ε, αλλά όλα αυτά θα προβλεφθούν στο πακέτο κινητικότητα. με την λεγόμενη ευρωβινιέτα. Όχι οικολογικό φόρο όπως κάποιοι φοβούνται. Ευρωβινιέτα είναι διαφορετικό. Και το τελευταίο ερώτημα που είναι ένα πραγματικό ερώτημα για το αυτόνομο όχημα. Είμαστε σε μια φάση ιδιαίτερη όπω είπατε, αλλά το αυτοκίνητο πηγαίνει μόνο του ήδη. Όχι. Ανταλλάσσουν πλήρω μεταξύ του τα οχήματα. Είναι ε, αλληλοσυνδεδεμένα. Σα λέει προσοχή στα 59 ε, έχει ε, ατύχημα και το καθεξής. Υπάρχει, υπάρχει το αυτόνομο όχημα. Ο κύριο Ερτούκ το είπε, το ημιαυτόματο όχημα φτάνει το 2021. Σε κάποιες ευθείες ο οδηγός δεν χρειάζεται καν να κουμπάει το τιμόνι. Και μετά το αυτόνομο όχημα, είναι αυτό που είπε ο κύριο Ερτούκ πολύ καλά, το θέμα της ευθύνη, το αυτόνομο όχημα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αν δεν ρυθμίσουμε το θέμα των δεδομένων. Ένα αυτόνομο όχημα δεν μπορεί να πηγαίνει σε ένα δρόμο εάν δεν έχει την πληροφορία το φανάρι πρόκειται να γίνει πράσινο. Άρα το θέμα των ανοιχτών δεδομένων, των ελεύθερων δεδομένων, θα είναι ουσιαστικά το καύσιμο του αυτόνομου οχήματο. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Βίνταν Φαντεγκάμπ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, όταν μιλάμε για κοινωνικό ντάμπινγκ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αλλιώ υπάρχει μια τάση να μιλάμε για διατάξεις εργασίας που δεν ταιριάζουν ακριβώς στο εθνικό σύστημα και να τις λέμε κοινωνικό dumping. Βλέπουμε ότι η εσωτερική αγορά 502 εκατομμύρια άνθρωποι πράγματι θεωρεί ότι υπάρχουν και κάποιες κοινωνικές πτυχές στην απελευθέρωση. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, κατόπιν πρότασης της ε, κυρίας Τάισεν είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία η οποία θα δει το τι γίνεται με τις κοινωνικές συνθήκες. Εγώ βεβαίως είμαι Ολλανδός και να σας πω ότι ε, είμαι έκπληκτος με τις γαλλικές διατάξεις ε, περί εργασίες. Είναι πολύ αυστηρές. Είχαμε τεράστια προβλήματα με τους πιλότους ε, της Air France KLM γιατί οι Γάλλοι πιλότοι είχαν πολύ αυστηρές συνθήκες εργασίας και οι Ολλανδοί πιλότοι πολύ πιο ευέλικτες. Οπότε δεν παραγνωρίζω το πρόβλημα, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ζούμε στο κομμάτι εκείνο του κόσμου με τις καλύτερες συνθήκες εργασίας του κόσμου αν δείτε τι γίνεται στις ΗΠΑ ταυτόχρονα βεβαίως το πρόβλημα δεν θα φύγει με τα λόγια και οπωσδήποτε θα το ξαναδούμε στο πακέτο κινητικότητας αλλά ε, με μια Γαλλία πιο ευέλικτη. Κύριε Νταλούντε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς υπάρχουν πολλά πλέον εκτήματα. Η ασφάλεια π.χ. μας λένε ότι τα αυτοκίνητα θα έχουν μεγαλύτερη ασφαλεία. Οι άνθρωποι πίνουν ενόπνευμα, κουράζονται, και τα γεωταχή ούτως ή άλλως ε, είναι ακίνητα το 70% του χρόνου. Θα χρειάζονται λοιπόν λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερες θέσεις πάρκινγκ, καλύτερη ποιότητα ζωής στις πόλεις. Ε, θα πρέπει να περιοριστεί γενικά ο χρόνος οδήγησης αυτοκινήτων, αλλά η τεχνολογία για τα αυτοκίνητα αυτά θα είναι έτοιμη πριν από την νομοθεσία. Παραδείγματο χάρη όταν ένα αυτοκίνητο πρέπει να επιλέξει ποιον θα αποφύγει σε περίπτωση δυστυχήματος. Έχουμε πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σκόχ, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση από την Γερμανία για την ομοθεσία που είπατε που είναι του 1968 έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και καιρό γιατί λέει εκεί πέρα πως πρέπει ανα πάσα στιγμή να έχει τον έλεγχο του οχήματος ο οδηγός. Έχουν βγει δηλαδή συστήματα το ABS και το ESP που παρεμβαίνουν και δεν έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος ο οδηγός έτσι. Και αυτή τη στιγμή συντάσω μία έκθεση όπου ζητάμε ακριβώς να υπάρξει ένα σύστημα το οποίο θα φρενάρει αυτομάτως εάν δει ένα πεζό ή ποδηλάτη. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε περαιτέρω την ε, συνθήκη της Βιέννης ε, αν θέμε να προχωρήσει η θα πρεπει λοιπον οδήγηση. Μετά υπήρχε η άλλη ερώτηση για τις τεχνικές αυτές διατάξεις στα αυτοκίνητα. Δεν είναι αυτός σκοπός. Απλά ενημερώνουν για την συμπεριφορά του οδηγού. Και αν σκεφτούμε τώρα α, ε, σημερινή κατάσταση όπου κάνω νόημα σε κάποιον πεζό να περάσει πρέπει να βρούμε νέα συστήματα ε, για να κάνουμε σήματα αλλά πρέπει εμείς να διαμορφώσουμε το πλαίσιο, να είμαστε ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία και να δούμε τι θα έρθει. Ευχαριστούμε κύριε Κόχ και τώρα περνάμε απευθείας στον επόμενο βασικό μας προσκεκλημένο, έναν από τους βασικούς επαΐοντες του θέματος. Είστε ε, υπεύθυνος της Φαμπρίκ της Κινητικότητας, ε, του εργαστηρίου αυτοκινητικότητας και έχετε πολύ καλή γνώση για να μας πείτε τι προβλέπετε για το μέλλον, τι ε, ετοιμάζετε και θα έχουμε κι άλλη συζήτηση, ε, διάλογο με τους πολίτες σε δεύτερη φάση. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Είμαι υπεύθυνο τη φαμπρίκ ε, τη κινητικότητα, τη ε, αυτού, αλλά σήμερα θέλω να μιλήσω για την προσωπική μου άποψη, για το ποιο θα μπορούσε να είναι, όχι ποιο θα έπρεπε να είναι το μέλλον τη κινητικότητα ε, μέσα σε λίγα χρόνια. Προσωπικώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε για την αστική κινητικότητα στο ποδήλατο. Αυτό είναι το μέλλον τη αστική κινητικότητα. Σήμερα όμω δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Θα μιλήσω για τι τάσει που αναλύουμε τα τελευταία χρόνια και οι οποίες επιταχύνονται αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι το θέμα της, ε, κοινων, της οικονομίας και πώς θέλουμε να μοιραστούμε τα ωφέλη της, είναι το θέμα της παραγωγής, είναι το θέμα των χρηστών. Γενιές. Είδαμε να υπάρχουν πολλές διαφορές τα τελευταία χρόνια στους νέους, στο επίπεδο των νέων. Επειδή οι νέες γενιές έχουν αλλάξει στις συμπεριφορέ τους, σε σχέση με το παρελθόν, έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Τι βλέπουμε λοιπόν, έρευνες στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή στην Ιαπωνία, όποτε ερωτούν το κοινό τι ήταν αυτό που θα θέλεις να ξεφορτωθείς από τα πράγματά σου, είναι, δεν θα ήθελα να ξεχάσω και να παρατήσω το smartphone τον απολογιστή μου ή το αυτοκίνητό μου. Ε, αυτό αλλάζει λίγο στις μεγαλύτερες γενιές Ας δούμε τι γίνεται με το δίπλωμα οδήγησης ε, λόγου χάρη. Βλέπετε, εσείς που ξέρετε από Βρυξέλλες την ηλικία που περνάει ο κόσμο στι εξετάσει για το δίπλωμα. Τι βλέπουμε. Κάθε δεκαετία, μόνο μέσα σε μια δεκαετία, οι γαλάζιε κολόνε δραστικά μειώνονται. Διότι ο κόσμο δεν έχει ανάγκη να οδηγεί ένα αυτοκίνητο μόλι γίνει 18. Αυτό το βλέπουμε παντού πλέον. Παντού ε, στι ανεπτυγμένε χώρε. Οι νέε γενιέ λοιπόν είναι ένα βασικό θέμα. Το άλλο είναι η κατανομή, η κοινή χρήση, το πώς μπορούμε να μοιραστούμε τα πράγματα. Αυτό το μοίρασμα μας οδηγεί στο μόνο μονόκερο στις ευρωπαϊκές μεταφορές, το, καρ, το μπλα μπλα καρ. Είναι ε, πραγματικά καινοτόμος η δική τους σύλληψη. έχουν καταφέρει να αποδείξουν ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τα μέλη του μπλα μπλα περισσότερο από τους συναδέλφους τους ή τις επαφές του Facebook. Αυτό θα πει ότι εντός του συστήματός τους είναι αξιόπιστη. Ο κόσμος είναι έτοιμος να επιβιβαστεί στο όχημα κάποιου που είναι εντελώς άγνωστος. Επειδή η πλατφόρμα είναι τόσο ισχυρή που πραγματικά μπορεί κανείς να εμπιστευτεί την πλατφόρμα. Αυτό που βλέπουμε είναι ε, μέσα από αυτές τις νέες πλατφόρμες, από αυτές τις νέες εφαρμογές, ότι υπάρχουν πολλά ε, συστήματα μοιράσματος της οδήγησης. Το βλέπετε στο Google με αυτές τις εφαρμογές, αλλά ξέρουμε και το Facebook προσφέρει τις ανάλογες. Αναπτύσσει αυτού του είδους τις επιλογές. Πολύ γρήγορα, διότι έχουν ε, το σχετικό πρόγραμμα. Εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον. Ε, η όλη ιδέα λοιπόν είναι να δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε με αυτές τις ιδέες μοιράσματο των αυτοκινήτων. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τους παραδοσιακού τρόπους οδήγησης. Και δεν τα έχουμε δει ακόμα όλα. Δεν σκεφτόταν κανείς τι αντίκτυπο θα έχει το BlaBlaCar ω νέο αφιχτή στην αγορά ε, των αυτοκινήτων και υπάρχει μεγάλο μοίρασμα των αυτοκινήτων πλέον. Είναι ένα σύστημα που υπήρχε από δεκαετίες, πάντοτε υπήρχε δυνατότητα να χρησιμοποιούν πάνω από δύο άνθρωποι το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά τώρα στα πλαίσια τη ανάπτυξη τη κινητικότητας, τη Γερμανία και το Βέλγιο βλέπουν να παίρνουν πολύ μεγάλε διαστάσει. Βλέπουμε λοιπόν αυτέ οι πλατφόρμε να ανθούν. Και αν κοιτάξει κανεί απλώ τι Βρυξέλλε, γιατί περισσότερο εδώ μένετε, μέσα σε ένα χρόνο γίναμε σχεδόν η πρωτεύουσα μοιράσματο αυτοκινήτων στην Ευρώπη για να μην πω στον κόσμο. Διότι όλοι οι οδηγοί αυτοκινήτων έχουν ε, χρησιμοποιήσει τέτοια πλατφόρμα. Επίσης, πέραν του μοιράσματο των αυτοκινήτων, μπορούν κι άλλοι να μοιραστούν τα αυτοκίνητα μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα από τη Λιόν για ένα Σαββατοκύριακο που υπάρχει μοίρασμα αυτοκινήτων μεταξύ πολλών διαφορετικών ανθρώπων. Όμω υπάρχει η ανάπτυξη και άλλων εναλλακτικών, όπως η ανάπτυξη των ε, μεγάλων διαδρομών λεωφορείων με μεγάλη άνθηση στη Γαλλία και τη Γερμανία. Ένα τρόπο να μοιραστεί κανεί τι εγκαταστάσει, τι υποδομέ, διότι στι αυτοκινητοδρόμου ε, έχουμε πολύ συχνά αυτοκίνητα και φορτηγά. Αλλά έχουμε πλέον και τα μακρών διαδρομών λεωφορεία. Ε, μέσα σε λίγα χρόνια μόνο αναπτύχθηκε ο τομέας αυτός με έναν μόνο μεγάλο ε, παράγοντα, μια μεγάλη εταιρεία που βασίζεται στα δεδομένα. Μπορούμε να μοιραστούμε κάθε είδου υποδομέ, όπω τη στάθμευση, το χώρο στάθμευση. Αυτή είναι μια ε, βαλγική εταιρεία, η και Υπάρχει μια αντίστοιχη στη Γαλλία, ε, ή αλλού στη Γερμανία, στο Μόναχο. Όλοι αυτοί βοηθούν του ε, του ιδιοκτήτε χώρων στάθμευση να εκμεταλλευτούν αυτούς τους χώρους στάθμευση όντω μια πόλη. Πέραν... Ναι, μπορείτε να προχωρήσετε. Ευχαριστώ. Μετά υπάρχει το θέμα της διαταραχής, της διακοπή. Πριν από τρία χρόνια είδαμε κάποιου από αυτού τους διαταράκτες να παίρνουν μεγάλη θέση στο όλο τοπίο και ε, πολλές φορές επιταχύνεται η δράση τους. έχετε ακούσει για τον Κάθα από τον προηγούμενο ομιλητή που δεν ήξερε τον καθά. Ξέρετε τι εννοούμε Google, Amazon και Facebook. Και Facebook. Ε, ευχαριστώ, αλλά αυτό θα μπορούσε κανείς να το αντιπαραθέσει στο ΝΑΤΟ. Ξέρει κανείς τι είναι το ΝΑΤΟ. Κανείς. Τους ξέρετε. Είναι το Netflix, το Airbnb, το Bloomberg και το Tesla. Όλα αυτά αναπτύσσονται πολύ γρηγορότερα από τον ΚΑΦΑ, διότι χρησιμοποιούν τον ΚΑΦΑ για να αναπτυχθούν. Η οικονομία πλατφόρμας μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν τι συμβαίνει με τα ΝΑΤΟ και τα ΓΚΑΦΑ. Είναι εταιρείε που αναγκάσαν την θέσπιση του πρώτου ε, ψηφιακού πρεσβευτή. Διότι πρέπει να συνεργαστεί μαζί τους αλλά και να τους ε, ε, δαμάσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί μεταβάλλονται διαρκώ και μεταμορφώνουν και τον τομέα των μεταφορών. Να τα τανάτου. Ε, ευχαριστώ, προχωρήστε. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το Uber, έχει γίνει τόσο πολύ κουβέντα γι' αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ίσω είναι καλό να υπάρχουν αυτοί οι παράγοντε διαταραχή διότι έχει γίνει πολλή κουβέντα για το μέλλον των Ευρωπαϊκών Μεταφορών σε αυτή την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα πράγματα δεν ε, κινούνται και πάρα πολύ γρήγορα. Σκεφτείτε τι συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο στι Βρυξέλλε. Στι Βρυξέλλε χρειάστηκε να κλείσει ένα ολόκληρο, ε, ένα, μια ολόκληρη διάβαση οδογέφυρα. Διότι δεν μπορούσε να βρεθεί λύση για ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Θα μπορούσαν πολλά να έχουν γίνει. Μια γραμμή λεωφορείου να ε, στηθεί. Κάτι ω προσωρινή λύση. Αλλά δεν έγινε και υπήρξε μια μεγάλη διαταραχή. Βεβαίω οι παράγοντε αυτοί λοιπόν διαταράσσουν τι ισορροπίε τοπικά με μια τοπική προσέγγιση. Και τέταρτη, το τέταρτο σημείο που θέλω να σταθώ είναι η διασύνδεση. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε αυτή τη γενιά τη ε, συμμετοχική οικονομία, των ε, παραγόντων, των παραγόντων που διαταράσσουν. Πρέπει να υπάρξει σωστή διασύνδεση. Ίσως με ίση μαχήριση η μεταχείριση ίσω με, το μοίρασμα των αυτοκινήτων, με τον εξορθολογισμό των τιμών. Πολλά πολλά πράγματα μπορεί να είναι μέρος αυτή της διασύνδεση. Όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι περισσότεροι φορεί που είναι πολύ καλά διασυνδεδεμένοι δεν είναι ευρωπαϊκοί. Google. Ένα δις χρήστες ε, καθημερινά χρησιμοποιούν το Google Maps. Οι ευρωπαϊκέ startup με αν είχαν τέτοιο ανάπτυξη θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν. Αυτό τώρα είναι τι έκανα χθε. Ε, η διαδρομή που έκανα χθε με το Google Maps. Δεν είναι ακριβώς ε, τα πάντα, αλλά το Google ξέρει πάρα πολλά για μένα. Ξέρει σε ποια εκδήλωση πήγα από το Ισραήλ, μετά που πήγα στους φίλους μου και που έμεινα εκεί ένα δίωρο. Ξέρει τα πάντα. Ξέρουν ότι πήρα το ποδήλατο για 2,5 χιλιόμετρα, ξέρουν ότι ε, σήμερα έπρεπε να έρθει εδώ, ξέρουν τα πάντα για το πρόγραμμά μου. Αυτό είναι λοιπόν η τέταρτη βασική λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Το άλλο είναι αυτό που πενήθηκα πριν από το λόγο μου. Μπορείτε να προχωρήσετε. Παρακάτω. Αυτοματοποίηση. Στη μέση ακριβώ τη γενιά αυτή τη ψηφιοποίηση με του παράγοντε διαταραχή και τα άλλα στοιχεία που ανέφερα, βλέπετε την αυτοματοποίηση. Αυτό θα μπορούσε να τα συμπεριλάβει όλα σε ένα σύστημα το οποίο δεν θα το κινούν οι δημόσιες αρχές, αλλά οι ιδιωτικοί φορείς σε συνεργασία μεταξύ τους. Διότι δεν είναι πλέον ε, έγκλημα. Ε, το Tesla μας δίνει τη δυνατότητα σε ένα smartphone με ένα νέο λογισμικό να βρούμε άλλη λύση για τη στάθμευση. Αυτό είναι ένα δίκτυο που έχει αναπτυχθεί. Και η Wimo θα προσφέρει υπηρεσίες οδήγησης ε, ήδη τον επόμενο μήνα στο Phoenix των ΗΠΑ βλέπουμε ότι είμαστε ακόμη στο επίπεδο 2 με την αυτοματοποίηση, αλλά πηγαίνουμε πολύ γρήγορα. Και τα πράγματα θα πάνε ακόμη πιο γρήγορα. Και τελευταίε κουβέντε για το νέο οικοσύστημα. Υπάρχει ένα παγκόσμιο πλέον οικοσύστημα, αλλά λείπει κάτι. Οι δημόσιοι προπολογισμοί δεν συμμετέχουν σε όλο αυτό το σύστημα. Υπάρχουν οι αυτοκινητοβιομηχανίε, οι πλατφόρμες, η αυτοματοποίηση και οι παραγοντές τη. οι σχετικές εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, η Google, η Apple, η Microsoft και ούτω καθεξής εδώ θα πρέπει να το ε, έχουμε υπόψη. Και μια κουβέντα για την κινητικότητα μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Η δική μας ε, εταιρεία, η Fabric Mobility, ε, το εργαστήριο κινητικότητας έχει ξεκινήσει στη Γαλλία πρόσφατα και καταφέραμε να κάνουμε τις εταιρείες startup την κινητικότητα να μην είναι μονοκερη Υπάρχουν startup που ενδιαφέρονται να δουν αυτό το οικοσύστημα. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιήσουμε και άλλα οικοσυστήματα της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και να συσχετιστούμε, να συνεργαστούμε μαζί τους. Οι εταιρείε startup δεν χρειάζονται μόνο χρήμα, χρειάζονται και στήριξη, πολιτική στήριξη, ε, καινοτόμα νομοθεσία. Ε, χρειάζονται πολλά. Βεβαίω χρειάζονται και το η χρηματοδότηση, αλλά δεν είναι αυτό αρκετό. Ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίαση. Αυτή η παρουσίαση που είναι άκρος ανησυχητική και μας δείχνει ότι οι νέες τεχνολογίες στην ουσία ε, μπορούν να αναχαιτήσουν τη τεχνολογία. Τι σημαίνει συνεργατική οικονομία. Ε, υφίσταται. Ε, εδώ σας μιλώ ως βουλευτής, δεν το πιστεύω τι μπορεί να γίνει με την συνεργατική οικονομία. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα νομικό κενό και εδώ τίθενται ουσιαστικά ερωτήματα. Ε, μιλήσαμε για διάφορες προκλήσεις, κλιματικές περιβάλλοντος. Ε, εγώ όμως θα ήθελα να ασχοληθούμε με το κοινωνικό ντάμπινγκ. Η κυρία Ρεβονταλόν γνωρίζει αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό θα της δώσω το λόγο γιατί ετέθηκε αυτό το ερώτημα και θα πρέπει να δοθεί μία απάντηση. Ευχαριστώ. Ίσως με αυτό τον, κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να, κάνουμε μια, να βρούμε μια εξισορρόπηση ως προς τις θέσεις μας. Αν δούμε τον τομέα των μεταφορών, βλέπουμε ότι δύο πόλοι είναι το περιβάλλον και τα κοινωνικά ζητήματα. Όπως ξέρετε, ως προς το κοινωνικό ντάμπινγκ υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό η Επιτροπή Απασχόλησης, όπως και η δική μας ε, Επιτροπή. Δεν συμμερίζομαι την άποψη του κυρίου Βαντεκάμπ. Ε, δεν πρόκειται για ανέλικτα σχήματα Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προασπίσουμε, να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους ε, ε, ως προς την απελευθέρωση. Αυτό είναι μια πολιτική άποψη. Και στο πακέτο της κινητικότητας υπάρχει μια κοινωνική πτυχή που θα πρέπει να ξαναδούμε. Και υπάρχει και ένα άλλο κείμενο, αναθεώρηση της οδηγίας των αποσπασμένων εργαζομένων όπου θεωρούμε ότι ο τομέας μεταφορών δεν θα πρέπει να μπει στην άκρη. Δηλαδή οι εργαζόμενοι στον τομέα μεταφορών να μην έχουν τα, ίδια δικαιώματα με τους άλλους ε, τομείς. Εκπροσωπούμε πολιτικές ομάδες και κινήματα, γι' αυτό έχουμε να κάνουμε και με διαφορετικές επιλογές. Δεν ξέχασα τους Τέλιτσκα και Κράμερ, αλλά υπάρχουν και άλλοι πολίτες που θα ήθελαν το λόγο και θα τους τον δώσουμε για να υποβάλουν τα ερωτήματά τους. Έχετε το λόγο. Εδώ θα βάλω ε, χρονόμετρο. Θα ήθελα να μιλήσω για την κινητικότητα η οποία μπορεί να ε, απασφαλίσει τα οικονομικά δικαιώματα και τι γίνεται ακριβώς όταν μιλάμε για την ιδιωτικότητα. Πώς όταν μεταβαίνουμε από το ένα σημείο στο άλλο ως προς την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Γι' αυτό πιστεύω ότι η κινητικότητα είναι ευάλωτη. Κάποιος άλλος που ζήτησε το λόγο. Ο κύριος με το πράσινο τουιντ. Θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ερώτημα που σχετίζεται με την αστική κινητικότητα αλλά και με την κοινωνική πτυχή του θέματος. Ως προς την δωρεάν παροχή υπηρεσιών γίνεται μια θεσμική συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ε, η ερώτησή μου είναι απλή. Τι πιστεύετε ως προς τις δωρεάν μεταφορές και ποιο είναι το μέλλον αυτής της ε, πορείας. Ο άλλος κύριος ε, ως προς το, τις δωρεάν μεταφορές θα ήθελα να πω ότι δεν αμφισβητούμε ότι ο σιδηρόδρομος είναι πιο ασφαλής σε σχέση με τις οδικές μεταφορές. Πιστεύω ότι εάν υπάρχει, υπάρχουν δωρεάν μεταφορές ως προς τη, τους σιδηροδρόμους θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την κινητικότητα. Επίσης θα γινόταν μεγαλύτερη χρήση των ε, μαζικών μέσων μεταφοράς γιατί έχουμε μία αύξηση 175% τη στιγμή που υπάρχει η δωρεάν παροχή ενώ στο Βέλγιο υπάρχει μείωση χρήσης κατά 16% άρα θα έχουμε περισσότερα ε, μάλλον λιγότερα οχήματα στους δρόμους αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό τη η χρηματοδότηση. Εγώ είμαι Βέλγος και ε, βασίζομαι... Ένα λεπτό μόνο. Διακόπτη πρόεδρος. Ε, αν λάβουμε υπόψη την SNCB θα έπρεπε να γίνει χρηματοδότηση ενός δις ε, αν γίνονται δωρεάν οι μεταφορές γιατί δεν θα χρειάζονταν ούτε ελεγκτές ούτε έκδοση εισιτηρίων. Άρα θα είχαμε εξοικονόμηση μισού δις. Εάν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει και συγχρηματοδότηση του βελγικού κράτους των οχημάτων μεγάλων εταιριών, μπορούμε να πούμε ότι αυτό το κόστος θα ε, συρρυκνωθεί και αυτό θα οδηγούσε σε μεγάλες εξοικονομίες. Είναι ο Γκαμπριέλ ε, και είμαι φοιτητή στο Παρίσι, θέλω να ε, μιλήσουμε για τον ομοιογενή χαρακτήρα καταβολής αντιτίμου μεταφορών, δηλαδή με ε, μία συνδρομή θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα μέσα στο Παρίσι, Βερολίνο ή η Μαδρίτη τη στιγμή που υπάρχει συνδεσιμότητα αυτών των πόλεων. Μπορούμε να προβάλλουμε αυτή την πλατφόρμα. Ε, είμαι φοιτήτρια στο Παρίσι και έχω την εντύπωση ότι μιλήσαμε είτε για τις σιδηροδρομικές είτε για τις οδικές μεταφορές. Ενώ ε, υπάρχει στο Παρίσι και ένας άλλος τρόπος μεταφορών οι ποτάμιες μεταφορές και αυτό αφορά τα εμπορεύματα αλλά και τους επιβάτες. Ποια είναι η δυνατότητα στις μεγάλες πόλεις με ποτάμια. Υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Η επόμενη ομιλήτρια. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Και εγώ σπουδάζω στο Παρίσι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρουσίαση για την διευκόλυνση των ε, μεταφορών. Ε, του μιλάμε για μπλαμπλακάρι, φλίξπας. Και αυτό γίνεται κυρίως βεβαίω ε, online. Αλλά υπάρχουν και κάποιες βελτιώσεις στον στις υποδομές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την κατάσταση. Για εμένα ως ε, νεαρή γυναίκα έχει σημασία και η ασφάλεια. Ε, θα μπορούσαν λοιπόν να έχουμε και κάποια ε, μέτρα φυσικά υποδομών. Σας ευχαριστώ. Ο νεαρός εκεί με το πουλόβερ το κόκκινο. Ευχαριστώ. Είχα και εγώ δύο ερωτήσει, αλλά τις έθεσαν οι προηγούμενοι. Θα τα πω γρήγορα. Τέλο πάντων, δεν είμαι συνηθισμένο να μιλάω στο κοινό και είναι και λίγο χρόνο. Ε, όταν λαμβάνουμε υπόψη ότι οι μεταφορέ έχουν, έχουν παίξει συγκεκριμένο ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία. Εγώ διαρωτώ με πότε θα υπάρξει μια φιλόδοξη πολιτική. Κρίμα που έφυγαν κάποιοι από του συναδέλφου σα. Αλλά μια φιλόδοξη πολιτική για το Interrail, το ευρωπαϊκό Interrail, όχι μόνο για του αεροδρόμου, αλλά και όλε τι μεταφορέ. Και η ερώτηση που μου φάνηκε κέρια είναι αυτή για την επισφάλεια. Υπάρχουν πολλέ ε, κοινωνικέ ανισότητε ακόμη, ε, κυρίω ε, ω προ την κινητικότητα. Μιλάμε για διαφορετικά μέσα μεταφορά, διαφορετικό τρόπο όπω να συμμετείχε κανεί μέσω των πλατφορμών συνεργασία και που πρέπει κανείς να πληρώνει. Δεν είναι το σύστημα το λογικό να πληρώνονται όλα, γιατί πιο επισφαλείς, αυτοί που γνωρίζουν μεγαλύτερη επισφάλεια, είναι αποκλεισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις. Το θέμα των δεδομένων. Το θέμα των δεδομένων που μας οδηγεί στο θέμα της κυβερνοασφάλειας. Μεγάλο ερώτημα, διότι Εάν μας ε, επιτεθεί κάποιος hacker θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η, λογική... αντίληψη ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας. Τώρα, για τις διαφορέ τη μεταφορές, διαφορέ τη επενδύση είναι ένα από του λόγου. Τα αυτοκίνητα υπηρεσίας, δεν ξέρω κατά πόσον είναι διαθέσιμα στο Βέλγιο. Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει αυτό, αλλά σωστά το είπατε και εσείς υπάρχει επισφάλεια στις μεταφορές. Ξέρουμε την ενεργειακή φτώχεια, άνθρωποι που δεν μπορούν να ζεσταθούν το χειμώνα και δεν μπορούν να πληρώσουν το ε, λογαριασμό τους κάθε μήνα, το λογαριασμό της θέρμανσης. Αυτό είναι επισφάλεια. Η επισφάλεια είναι φτώχεια, φτώχεια στις μεταφορές. Ε, στη Γαλλία εκτιμάμε σε 8 εκατομμύρια τα άτομα που είναι φτωχά ω προ τι μεταφορές. Τι θα πει αυτό. Θα πει ανθρωποί που δεν έχουν πρόσβαση στις μεταφορές. Ε, δεν καλύπτεται η περιοχή τους ή η τιμή τη μεταφορά, της μεταφοράς είναι πολύ υψηλή αυτός που δεν, είναι, που δεν έχει δυνατότητα κινητικότητα που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, αποκλείται από τον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί υπάρχει ρήγμα, κοινωνική ρήξη. Δεν είναι εδαφική ή γεωγραφική ή τοπογραφική, είναι κοινωνική ανισότητα, όπως μιλάμε για την ψηφιακή ανισότητα. Μπορεί να μιλάμε για το αυτόνομο όχημα, όμως από αύριο μπορεί να δημιουργήσει πραγματική ρήξη. Ε, Δηλαδή θα είναι οι νέοι των πόλεων που θα είναι και συνδεδεμένοι παντού και αυτοί που ζουν ε, στην Ήπεθρο και δεν, ξέρουν, ε, δεν έχουν πουθενά πρόσβαση. Είναι λοιπόν ένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν μπορώ βεβαίω να απαντήσω σε όλα εγώ, διότι κανεί δεν μου μετράει το δικό μου χρόνο ομιλία. Θα ζητήσω λοιπόν από του συναδέλφου να πάρουν το λόγο και να πούν και αυτοί το δικό του. Κύριε Βαντενκάμπ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε πέντε σημεία. Πρώτα απ' όλα η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να λάβει συγχαρητήρια γιατί προστατεύουμε την ιδιωτική ζωή στον σχετικό κανονισμό μετά από πολύ εκτεταμένες συζητήσεις αλλά εδώ πέρα θα συμφωνήσω με τον κύριο Τακούνε αν το λέω σωστά το όνομα ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις πάνε τόσο γρήγορα ώστε η προστασία της ιδιωτικής ζωής μένει πίσω κάποια στιγμή. Το δεύτερο. Πρέπει να προσέξουμε να μην, δώσουμε, να μην δίνουμε μόνοι μας τα πάντα στην Google και μετά να λέμε «Α, ναι, αλλά δεν προστατεύεται την ιδιωτική μας ζωή». Ε, το βλέπετε με τα ποδήλατα στις πόλεις των Βρυξελών αλλά βλέπετε ότι πολλά τα δίνουμε μόνοι μας λοιπόν κύρια Πρόεδρε για τις ε, δημόσιες συγκοινωνίες νομίζω ότι ο Πρόεδρος Μακρόν είναι ο αρμόδιος εδώ εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις συγκοινωνίες δωρεάν για όλους ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η δικιά μας δουλειά αυτό ανήκει στη λεγόμενη επικουρικότητα και ξέρω πως και η Δήμαρχος των Παρισίων είναι μια πολύ μοντέρνα γυναίκα και νομίζω ότι αυτό είναι ούτως ή άλλως εκτός αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναφερθώ λίγο στη συμπατριώτησά μου που είπε ότι θέλω να έχω κάποιο φυσικό περιβάλλον που θα με κάνει να νιώθω ασφαλής ε, τη νύχτα, το βράδυ όταν είμαι μόνη. Αυτά ε, είναι θέμα αρμοδιότητας ε, Δήμου Παρισίων. Και να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω αν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι. Το Interrail είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Βεβαίως κάτι ε, το επίμαχο στην Ολλανδία γιατί στην Ολλανδία θεωρούν ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ήδη που είναι δωρεάν ε, βεβαίως ο Μάνφετ Βέμπερ ο πρόεδρος μας είχε προτείνει κάθε 18χρονος να έχει ένα ειστήριο για 15 μέρες για την Ευρώπη αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ Κύριε Φαντεκάμ, κύριε Τενίτσικα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ δεν βλέπω κάποια πολιτική ομάδα εντός του Κοινοβουλίου που να είναι κατά των κοινωνικών δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποια μέσα μεταφοράς υπάρχουν εταιρείε ή άτομα που κάνουν κατάχρηση της νομοθεσίας. Α, είναι θέμα μετά εθνικών αρχών να εφαρμόσουν την νομοθεσία. Απ' την άλλη, αυτό το οποίο βλέπουμε ε, στο κοινωνικό dumping ε, είναι ουσιαστικά προστατευτισμός και υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της εσωτερικής αγοράς και τα κράτη-μέλη λαμβάνουν μεμονωμένα μέτρα που έχουν τεράστιες συνέπειες για την εσωτερική αγορά και για εμάς ως καταναλωτές. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, δωρεάν ε, δημόσιες μεταφορές. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φαντεκαμπ. Αν θέλει κάποια χώρα να το κάνει, καλώς. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είτε χρειώνεστε είτε όχι, θα το πληρώσετε μέσω φόρων, ε, αν είναι δωρεάν. Ε, και, και σε... Βεβαίω υπάρχει και το δημόσιο χρέο. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να φροντίσουμε κάποιες από τις πιο περιβαλλοντικά φιλικές ε, μορφές μεταφορών ε, να απελευθερωθούν από δέσμα οπωσδήποτε. Τέλος μιλάμε για περιβάλλον, ε, κοινωνικά ζητήματα κτλ. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και αυτό ήταν στην έκθεσή μου για την αεροπορία ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης συνδεσιμότητας που θα διασφαλίζει ότι θα έχουμε διασύνδεση για τα άτομα, για τους πολίτες, ε, τους ε, πελάτες και είμαι σίγουρο ότι αυτός ο δείκτης ε, θα γίνει πραγματικότητα πολύ σύντομα. Κύριος Κράμερ, γρήγορα για ένα λεπτό. Ναι, το, αναφέρθηκε το software του Diesel. Πράγματι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή ρύθμιση, μια εξέταση ε, γιατί οι χώρες απέτυχαν να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε, οπότε χρειάζεται ευρωπαϊκός έλεγχος. Κοινωνικό dumping. Είχαμε οδηγό Ρουμάνο που οδηγούσε επί 8 μήνες Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία και κοιμόταν μόνο στο αυτοκίνητό του και πληρωνόταν κάτω από 300 ευρώ. Αυτή είναι σύγχρονη σκλαβιά. Πρέπει να δούμε τον ταχογράφο, να δούμε πού πάει, αν αυτός ο άνθρωπος είναι τον περισσότερο χρόνο στη Γερμανία να πληρώνεται γερμανικό μισθό, όχι ρουμάνικο. Δωρεάν μεταφορές. Δωρεάν δεν υπάρχει. Κάποιος το πληρώνει. Για μαθητές, φοιτητές, για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να το πληρώσουν πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ε, γιατί είναι πράγματι βάση για τη ζωή. Αλλά κοιτάξτε, εγώ είμαι από την ε, Γερμανία. Αν κόβαμε το 18 cent του ευρώ που επιδοτείται το ντίζελ θα μπορούσαμε να το χρηματοδοτήσουμε. Και βεβαίως ε, έχει μεγάλη σημασία και η προστασία των δεδομένων. Πρέπει να έχουμε δίκαιο ανταγωνισμό. Πρέπει δηλαδή να στηρίξουμε τους σιδηρόδρομους. Ε, αλλά τι κάνουμε στην Ευρώπη, στηρίζουμε τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι λάθος και πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστούμε κύριε Κράμερ. Ο κύριος Κόρ. Ευχαριστώ. Ναι, από το Παρίσι ε, ήρθε η πρόταση να υπάρχει η δυνατότητα να πάει κανείς από πόρτα σε πόρτα με ένα μόνο ειστήριο. Κάτι με το οποίο συμφωνώ πλήρως. Επίσης, ε, να υπάρχει η δυνατότητα πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για το τι γίνεται για όλα τα μέσα μεταφορά και να ε, ειστήριο το οποίο θα αφορά διαφορετικά μέσα μεταφοράς από το ταξί, στο σιδηροδρομικό σταθμό, στο αεροπλάνο κτλ. Και είπαμε ότι εάν δεν γίνει κάτι μέχρι το 2020 από τις επιχειρήσεις θα περάσουμε εμείς νόμο. Ε, τα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο δεν είναι ακόμα τόσο ικανοποιητικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος γύρος ερωτήσεων και μετά θα περάσουμε στα κοινωνικά δίκτυα και θα δοθούν απαντήσεις και ο εμπειρογνώμονάς μας θα απαντήσει στις ε, ερωτήσεις περί ατέλειας, εδαφικού κατακαιρματισμού και ούτω καθεξής. Ερωτήσεις παρακαλώ. Συγγνώμη που ξαναπαρεμβαίνω αλλά μετά από όσα ελέγχθησαν πρέπει να το κάνω. Κατηγορείται τα κράτη όταν ξέρουμε ότι η Γαλλία και η Γερμανία ζητούν να υπάρχουν οι ίδιοι μισθοί για τους οδηγούς ε, που διανύουν τη Γερμανία και τη Γαλλία, ενώ η Κομισιόν προσπαθεί να θέσει προσκόμματα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί και εσείς είσαστε υπεύθυνοι, όχι μόνο τα κράτη, μην τα ρίχνετε στα κράτη. Ως προς την ατέλεια, θα ήθελα να μιλήσουμε για κοινωνικό αντίτιμο και συμφωνώ για μία φορά με τον κύριο Κράμερ. Θα πρέπει οι φοιτητέ να μπορούν δωρεάν να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στις δημόσιες μεταφορές, με συγχωρείτε. γιατί θα πρέπει να τους γίνει συνήθεια να χρησιμοποιούν τα μασίκα μεταφοράς. Ως προς τις πλατφόρμες αποκλίνουν από όλους τους κανόνες γιατί είναι διεθνείς, δεν φέρουν καμία ευθύνη ως προς την απασχολησιμότητα και οι μισθωτοί θεωρούνται ε, επιχειρηματίε. Λυπάμαι, ε, κύριε Βαντερκάμπ, θα ήθελα, που δεν είσαστε εδώ, θα ήθελα ε, εσείς να μοιραστείτε τη ζωή ενός φτωχού τουλάχιστον για μισή μέρα. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Είμαι ο Αλφόν, σπουδάζω οικονομία και βλέπω ότι στις κουβέντε μα μιλάμε για τα αυτοκίνητα και τι λύσει των δημόσιων συγκοινωνιών για να αντιμετωπίσουμε το κυκλοφορικό στην Ευρώπη και να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου. Ε, εδώ λοιπόν σε σχέση με τι δημόσιε υπηρεσίε θέλω να μιλήσω για την Επιτροπή και τι προτάσει τη για τι πόλει. Διότι υπάρχουν αυτοκίνητα ε, που ρηπαίνουν πάρα πολύ στα κέντρα των πόλεων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο κέντρο τη πόλη. Στο Παρίσι το 2016 έχει προβλεφθεί διαφορετική ε, επιβολή τελών και ε, στη Γερμανία σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες πόλεις και υπάρχουν γειτονιές όπου υπάρχουν συγκεκριμένα ωράρια με συγκεκριμένα αυτοκίνητα που επιτρέπονται ή όχι. Μήπως έπρεπε λοιπόν να γίνει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική αυτή αντί να αφήσουμε τα διάφορα κράτη να τα αποφασίζουν μόνα τους ε, και συγκεκριμένα πολλέ φορέ οι ίδιοι οι Δήμοι. Μήπω πρέπει να ε, προβλέψουμε νέα κριτήρια ώστε να ελέγχουμε τα αυτοκίνητα και να ρυθμίσουμε τι δημόσιε κοινωνίε που ρηπαίνουν πάρα πολύ και που από ό,τι φαίνεται ε, θα τις χρησιμοποιήσει ο πληθυσμό αν ελέγχονται σωστά. Αλλιώ θα τα αφήσουμε στα χέρια των πόλων και ο καθένα θα κάνει ό,τι του κατεβαίνει, ενώ πρόκειται για το ίδιο θέμα στην ουσία. Ευχαριστούμε πολύ, Αλφόν. Μετά εκεί πίσω ναι, θα ξαναπάρω το λόγο για να δώσω μια μαρτυρία για τις πλατφόρμες συνεργασίες, τις πλατφόρμες μοιράσματος. Είναι ένα στοιχείο που θα υπάρξει στη νέα εκδοχή τη δική μα πλατφόρμα. Δεν κάνω εδώ τον εκπρόσωπο όλων των ποδηλατών, όλων των μπάκερ, αλλά όλου του χρήστε, του ε, ενθαρρύνουμε να μην ε, βλέπουν τον εαυτό τους, να μην παρουσιάζονται στους υπόλοιπους ως ε, απλώς εκμεταλλευτές της κατάστασης. Θέλουμε να δημιουργηθεί μια νέα εκδοχή, όπως είπαμε, να υπάρχουν μεν λύσεις ε, δωρεάν, αλλά υπάρχουν και αμοιβόμενες υπηρεσίες μην το δούμε με την προοπτική τη μετασοβιετική όπου τα πάντα προσφέρονται δωρεάν ε, ως δημόσια υπηρεσία σε αντίθεση με έναν καλπάζοντα ξέφρενο καπιταλισμό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά να μην ξεχνάμε την άλλη όψη του νομίσματος. Ε, με συγχωρείτε, αλλά πολύ γρήγορα. Ναι, ως προς την καινοτομία Υπάρχει η νοφιλελευθερία άποψη όπου η αγορά μαγικά έρχεται να ρυθμίσει μόνη της τα πάντα. Ως προς την κοινοτομία όμως, αρχικά χρειάζονται πολλά πράγματα. Χρήμα κυρίως, γιατί εντάξει ταλέντα, ιδέες, ε, εφευρετικότητα, ναι, αλλά κυρίως χρήμα. Ευχαριστώ πίσω σας. Ναι, να επανέλθω για ένα δευτερόλεπτο στο θέμα τη εδαφική ε, ρήξη του χάσματο που αναφέρθηκε προηγουμένω. Πρέπει να δούμε τι μεταφορέ από τη σκοπιά τη τεχνολογία και τη οικονομία μεν, αλλά δεν σκεφτήκαμε την πολεοδομία και τη χωροταξική μα διοργάνωση. Εάν θέλουμε ένα πρόγραμμα κινητικότητα, δεν, δεν πρέπει να ξεχνάμε να εξετάζουμε διαρκώ και επίμονα το, την διοργάνωσή μας στην χωροταξική. Ήδη από τη δεκαετία του 90 στη Γαλλία υπήρχε μια τέτοια πολυδημική πολιτική λόγου χάρη με τα απαραίτητα μέσα και αν δείτε τι έχει παραμείνει σήμερα σε σχέση με την ε, παραγωγή μεσοπόθεσμα και μακροπόθεσμα καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει τέτοια μετατόπιση και η κινητικότητα έχει διπλασιαστεί. Χρειάζεται καλύτερη εξισορρόπηση χωροταξικά. Ευχαριστούμε. Κύριε εκεί, στο βάθος, στο αριστερό μέρος της αίθουσας, από μένα. Α, δεν θέλατε το λόγο. Απλώς χαιρετούσατε. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα και πάλι. Η ερώτησή μου είναι λίγο κοινωνικού χαρακτήρα διότι μιλάμε για τις μεταφορές που θα πρέπει να είναι δωρεάν για να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες. Εδώ έχει ξαναρχίσει μια ολόκληρη συζήτηση στι εφημερίδε και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Η σεξουαλική παρενόχληση στι δημόσιε συγκοινωνίε. Διότι ξέρουμε ότι στατιστικέ μελέτε πρόσφατα δείχνουν ότι 100% των γυναικών λένε ότι έχουν δεχτεί παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση ή τέλο πάντων έχουν υπάρξει απόπειρε ασέλγια εναντίον τη δημόσια συγκοινωνία. Μάλιστα, δείχνουν οι μελέτε ότι μετά τι 2 το πρωί οι γυναίκε έχουν την τάση να παίρνουν ταξί για να επιστρέψουν σπίτι του παρά να παίρνουν τα δημόσια μέσα. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Πώ θα αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτή τη μάστιγα και κυρίω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι νομίζω το θέμα αυτό δεν απασχολεί μόνο την Γαλλία, αλλά όλε τι χώρε τη Ευρώπη Ευχαριστούμε. Άντε, μια τελευταία. Τελευταία όμως. Παρακαλώ. Γεια σας. Είμαι η Σαμπρίνα. Και εργάζομαι στην Ομοσπονδία για τα θύματα τροχαίων και ομαδικών ατυχημάτων. Πρέπει να σκεφτούμε στην Ευρώπη τι γίνεται όταν υπάρχει στις δημόσιες συγκοινωνίες ένα ατύχημα. Χρειάζεται εδώ μια εναρμόνιση ή θα εξετάζεται πάντα η κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Μήπω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να τα εναρμονίσει όλα αυτά για να υπάρχει συμμεταχειρήση των θυμάτων ασχέτω τη εθνικότητά του όταν υπάρχει ένα ατύχημα που αφορά πολλά άτομα ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πολύ. Τι ερωτήσει των κοινωνικών δικτύων τώρα. Από τα κοινωνικά δίκτυα έχουμε ακόμη πολλέ ερωτήσει που φτάνουν και δεν θα μπορέσουμε να τι καλύψουμε, δεν θα μπορέσουμε να τι θέσουμε όλε. Το δεύτερο θέμα που αναφέρθηκε ήταν δημόσια συγκοινωνίε. Με τον ε, Λοζέ Μπέιξ, ένα ανώνυμο μάλλον τον ε, χρήστη που από το Παρίσι που λέει ότι η κάρτα μου επιτρέπει να παίρνω το μετρό και το ποδήλατο, αλλά γιατί όχι όλους τους τρόπους μεταφορή. Ε, επίσης, ε, μια Αγγλίδα χρήστη μου λέει ε, ότι είχαμε ε, σχολικά λεωφορεία όταν μεγάλωνα, ηλεκτρικά να γίνουν, ηλεκτροκίνητα όλα, καθαρέ μεταφορέ για τα παιδιά και επίσης ένας άλλος Άγγλος χρήστη που μας λέει πότε σκοπεύετε να προβλέψετε ένα πάσο για όλα τα μέσα μεταφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης το οικουμενικό πάσο, ε, μετρό, ποδήλατο και όλοι, όλα τα άλλα μέσα μεταφορέ. και επίσης καθαρότερε δημόσιε κοινωνίε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολλέ ερωτήσει. Μιλάμε για τη μόλυνση στις πόλεις. Θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν μιλάμε για ε, πολιτική στα αστικά κέντρα, επειδή θα ασχοληθώ με την ευρωπαϊκή κινητικότητα στα αστικά κέντρα, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη ή στις πόλεις ορισμένους στόχους. Δεν είναι δυνατόν αυτό, γιατί δεν είναι θέμα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και ορισμένοι τομείς ε, παραμένουν ε, στο κεφάλαιο της επικουρικότητας. Δηλαδή ε, είναι κρατικής αρμοδιότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα. Θέτουμε στόχους ως προς την πολιτική στα αστικά κέντρα θα έχουμε μία δήλωση που θα που υπογράφει από τους Υπουργούς Μεταφορών εδώ και ένα χρόνο που μιλά για ενίσχυση της θέσης του ποδηλάτου στις πόλεις, δηλαδή ποδηλατόδρομους και ούτω καθεξής. Και τότε ο κύριος Κράμερ ήταν πρόεδρος της Επιτροπής. Όλοι μιλήσαμε για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου στα αστικά κέντρα. Τώρα αυτό θα πρέπει να το μεταφέρουν τα κράτη και οι πόλεις και να το κάνουν απτή πραγματικότητα. Πολλές φορές πρέπει να οχλούμε την Επιτροπή για να έχουμε αποτελέσματα και πολλές φορές το κάνουμε καλά. Ως προς την μόλυνση, αυτή είναι, είναι η πρόκληση του 21ου αιώνα. Ο Πόη λέει ότι η ασθένεια του 21ου αιώνα είναι η μόλυνση. Μιλάμε για 400.000 θανάτους, πρόωρους θανάτους εξαιτίας του ντίζελ. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ασχολούμαστε με την αντιμετώπιση της μόλυνσης, όχι μέσω μικρών στόχων. Θα πρέπει κάθε χώρα να έχει εθνική πολιτική για ανανασχέση τη μόλυνση και ξέρω ότι και στη Γαλλία ισχύει κάτι τέτοιο και θα ληφθούν υπόψη, θα ληφθεί υπόψη αυτός, αυτό το ζήτημα, η αντιμετώπιση μάλλον αυτής της ε, μάστιγας. Ως προς το εδαφικό που είναι θέμα ουσίας Δηλαδή δυστυχώς οι μεταφορές δεν ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Τώρα, ως προς την ε, σεξουαλική παρενόχληση στις δημόσιες μεταφορές, αυτό είναι θέμα ουσίας και ξέρω ότι η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών ασχολείται με αυτό το θέμα. Ίσως θα μπορούσαμε να προβάλλουμε μια συνεργασία και για το καθολικό πάσο και αυτό είναι θέμα αρμοδιότητας Επιτροπής Μεταφορών, δηλαδή περισσότερες ε, δημόσιες μεταφορές και μοίρασμα ε, μεταφορών και μετάβασης. Αυτό είναι ένας από τους μεγάλους στόχους μέσα στα πλαίσια της εναρμόνισης του ticketing. Έχουμε τον εμπειρογνώμονά μας εδώ και θα ήθελα να τον ρωτήσω τι σκέφτεται για αυτές τις προκλήσεις. Δεν μιλήσαμε για τις ποτάμιες μεταφορές ιδιαίτερα. Θα ήθελα όμως να τον ρωτήσω πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις εργασίες μας για την επαύριον. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι πιο σημαντικές προκλήσεις αναφέρθηκαν. Βεβαίω είναι πολύ επίγον να αντιμετωπίσουμε. Για τα δεδομένα και την ιδιωτικότητα είναι μεγάλη η μάχη, όχι μόνο για τις μεταφορές. Βεβαίω για τα άτομα. Αλλά το θέμα των δεδομένων είναι να αντιληφθούμε ότι οι εταιρείε αυτές έχουν τόσα δεδομένα πολύ περισσότερα από όλες τις εταιρείε δημοσίων μεταφορών. Η Google ξέρει πόσοι, σταθμοί, άνθρωποι βρίσκονται να πάει στιγμή σε ένα σταθμό στις Βρυξέλλες, το Παρίσι ή το Μάντσεστερ. Ε. Εάν έχουμε δεδομένα μπορούμε να κάνουμε τις μεταφορές να λειτουργούν πολύ πιο αποτελεσματικά. Αυτή είναι η μάχη. Μόλις έχουμε μπει στον πόλεμο της κινητικότητας. Ένας πραγματικός πόλεμος γιατί ε, η προηγούμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία έλεγε ότι ναι, να μειώσουμε τη μείωση των γιοταχή. Η μάχη δεν είναι πλέον ίδια. Βεβαίως να μειωθεί η χρήση των γιοταχή, αλλά πρέπει να μπορούμε και να ρυθμίσουμε όλους αυτούς τους νέους παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι. Κάθε μέρα έχουμε νέες υπηρεσίες ποδηλάτων, πράγματα όπως το Flexibus. Είναι σαν αστείο, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάει αυτό το Interrail για τους νέους εδώ και δύο χρόνια και το Flexibus θα ξεκινήσει σε δύο χρόνια. Interflex, 99 ευρώ ταξιδεύεις ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν Εντάξει, για μια λογική τιμή. Πρέπει να ε, κινητοποιηθούμε κι εμείς. Και υπάρχει μια σαφής ε, σύνδεση μεταξύ των δωρεάν μεταφορών. Ε, εγώ με κατά, δεν υπάρχει δωρεάν μεταφορές, νερά λοιπά. Δεν υπάρχουν ενέργεια. Έχουμε την περίπτωση στο Βέλγιο. Οι περισσότεροι μισθωτοί δεν πληρώνουν, Τους τα δίνουν συνήθω οι εταιρείε. 80% εταιρείε και 20% το κράτος. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, και ερχόμαστε εδώ πέρα στην πολεοδομία. Για τον λόγο αυτό ο κόσμος ζει εκτός Βρυξελών, 100 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες και δεν πληρώνουν τίποτα για να έρχονται κάθε μέρα στη δουλειά τους. Οπότε βεβαίως ε, η κοινωνική ένταξη είναι κάτι το κοινωνικό και πρέπει να υπάρχει κοινωνικό τιμολόγιο αλλά δωρεάν μεταφορές δεν είναι η λύση. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αλλά αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον ε, όσον αφορά τα ενιαία εισιτήρια λοιπά ε, με την μαζική κινητικότητα είναι ότι τι είναι μαζική κινητικότητα ένα πακέτο όπως έχουμε δηλαδή κινητό, ίντερνετ ε, κτλ σε ένα πακέτο 40-50 ευρώ και τηλεόραση, ε, το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα. Θα έχουμε ένα Netflix των ε, μεταφορών, π.χ. 150-200 ε, ευρώ για όλες τις υπηρεσίες. Βεβαίως δεν τις χρειάζεσαι όλες, γιατί μπορείς να πάρεις το τρένο 10 φορές το μήνα, να χρησιμοποιήσεις μια υπηρεσία αυτοκινήτων λίγες φορές τη βδομάδα για τέτοια πράγματα. Και ακριβώς αυτό το ενιαίο εισιτήριο πραγματικά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε τις περιπτώσεις στο Ελσίνκι Και ξεβλέπετε τι... Και βλέπετε ένα 13% του προϋπολογισμού ενός ε, σπιτιού πάει για την κινητικότητα. Αλλά από το 13% το 99% είναι για τα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητο και καύσιμα. Οπότε, εάν αναπτύξουμε ένα μαζικό πακέτο και έχουμε μία μάζα ανθρώπων που θα σταματήσει να έχει αυτοκίνητο και θα έχει εναλλακτικέ π.χ. Ε, κοινή χρήση αυτοκινήτων, θα έχουμε πολλά λεφτά για να έχουμε ένα κοινωνικό τιμολόγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί πολίτες, Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας κατά 15 λεπτά σε αυτή την εκδήλωση και θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Έχετε δύο επιλογές, είτε να μείνετε μαζί μας, είτε να... Α, θα μείνετε, θα μείνει θαύμα. Δεν σας λέω τη δεύτερη επιλογή. Τώρα θα δείτε μία πραγματική συνεδρίαση εργασίας. Δεν θα μπορείτε να υποβάλλετε όμως ερωτήσεις θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς θα γίνει. Στην Επιτροπή Μεταφορών υπάρχει, υπάρχουν διάφορα θέματα και εισηγητές. Θα ασχοληθούμε με το επόμενο θέμα που αφορά την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμου των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Για κάθε έκθεση υπάρχει, υπάρχει Άρα ο Νίκολα Καπούτο, ο εισηγητής μας, θα μας πει πού βρισκόμαστε. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία η πρόταση κανονισμού για την παρακολούθηση των στοιχείων και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στα βαρέα οχήματα θα είναι άλλη μία ψηφίδα ε, για να αναθεωρήσουμε αυτό το πλαίσιο εργασίας έτσι ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί με βάση τις ε, κλιματικές αλλαγές. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το σύστημα VECTO, το οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί για να ξέρουμε ε, την πραγματική κατανάλωση και τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Άρα έχει σημασία να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων και ως προς την βιωσιμότητα του πλαισίου. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να επιλέξουμε τα οχήματα αυτά για εντατική εκμετάλλευση. Θέλουμε λοιπόν να εξισορροπήσουμε τα στοιχεία αυτά και να αποφύγουμε αθέμητο ανταγωνισμό, βιομηχανική κατασκοπία ή οτιδήποτε άλλο που αφορά διάδοση ευαίσθητων στοιχείων θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα ε, ευαίσθητα στοιχεία και τα στοιχεία που να μπορούν να είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα. Τα ευαίσθητα στοιχεία δεν θα πρέπει να διαδοθούν. Δηλαδή μιλάμε για τον αριθμό της πινακίδας, ενώ τα στοιχεία που έχουν εμπορική σημασία και επιπτώσεις, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλες τις επιχειρήσεις πέρα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Σχετίζονται με τα στοιχεία ε, μετάδοσης, ελαστικά και ούτω καθεξής έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να μην μπορούν να έχουν ε, σχετικό πλεονέκτημα όπως ορίζουν οι συνθήκες στο άρθρο 81 και 82. Με ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε να εξισορροπήσουμε όλα τα συμφέροντα και να θέσουμε τις βάσεις πραγματικής ε, βιωσιμότητας για τους ε, φορείς, οικονομικούς φορείς. Περιμένω τις δικές σας υποδείξεις για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με το πακέτο της κινητικότητας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καπούτο. Βλέπω ότι πολλοί πολίτες αποχωρούν σιγά σιγά, όχι επειδή το θέμα δεν είναι ενδιαφέρον. αλλά ίσως ε, έχουν άλλα πράγματα να κάνουν. Σας ευχαριστώ, τους ευχαριστώ, είσαστε ευπρόσδεκτοι στην ε, Επιτροπή μας. Αυτή η εκδήλωση έγινε για πρώτη φορά, αλλά ίσως ε, να υπάρξουν και μεταγενέστερες. Εσείς θα σχεδιάσετε τις αυριανές πόλεις, πόλεις που θα πρέπει να είναι ανθεκτικές, ε, να έχουν βιωσιμότητα και μεταφορές πέρα από τα ζητήματα στέγης που υπάρχουν στις μεγάλες και μικρότερες πόλεις. Ένα χειροκρότημα για τους πολίτες μας. Ε, θα συνεχίσουμε την έκθεση Καπούτο και δίνω το λόγο στους συνεισηγητές. Βιρκούνεν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους Ευρωπαίους πολίτες που ήρθαν εδώ. Βλέπουμε εδώ πέρα πως έχουμε την έκθεση για τις εκπομπές δεξίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων και των εμβαρένων επαγγελματικών οχημάτων. Μιλάμε για τη μείωση του άνθρακα στι μεταφορέ. Ε, τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή μέχρι στιγμή είχαν ε, φέρει το μεγαλύτερο βάρο και τώρα θα καλυφθούν και τα βαρέα φορτηγά. Και βεβαίως ο στόχος εδώ πέρα είναι ακριβώς να δημιουργηθεί μια διαφάνεια στην αγορά Επίσης είναι σημαντικό τα βαρέα οχήματα να μπορούν και οι εταιρείες να μπορούν να συγκρίνουν τα πιο αποτελεσματικά οχήματα και βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα να προωθηθούν έτσι και νέες προδιαγραφές και αποτελεσματικότερα οχήματα και σημαντικό είναι να σημειώσουμε πως θα πρέπει ακριβώς να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις δυνατότητες των οχημάτων που επιστρέφουν και οχήματα τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία με την μία. Έτσι θα μειωθεί το κόστος των μεταφορών και οι εκπομπές. Οπότε τα μέλη αυτά τα οποία είχαν στη Φιλανδία πριν από λίγα χρόνια ε, θα θυμάστε ότι είδαμε και τα οικολογικά φορτηγά της Φιλανδίας και ακριβώς ε, ταξίδευαν σε πολύ μεγάλες ε, αποστάσεις. Και βεβαίως Πρέπει να δούμε και τις ε, πληροφορίες αυτές οι οποίες θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν αλλά θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ιδιωτικότητα είτε μιλάμε για την προσωπική ζωή είτε για λόγους ανταγωνισμού. Αυτά ευχαριστώ τον εισηγητή και αναμένω να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστούμε την κυρία ε, Βιρκίνεν, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι εκπομπές διοξιδίου του ανθράκα από βαρέα οχήματα που αποτελούν το 25% των εκπομπών του τομέα των μεταφορών. Γι' αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσουμε το όλο ζήτημα και τα στοιχεία να είναι συγκρίσιμα σύμφωνα με τον κανονισμό που προτείνεται είναι σαφές ότι όλοι οι συνομιλητές θα πρέπει να παραχωρήσουν στοιχεία, στοιχεία τα οποία η Επιτροπή θα μπορέσει να μελετήσει. Γι' αυτό τάσομαι υπέρ αυτής της ε, πρότασης, καθώς και της πρότασης του εισηγητή, που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, περάσει σε ε, κατεξουδότηση πράξης και όχι εκτελεστικές. Θα πρέπει να μειωθούν ορισμένα όρια που υπάρχουν ως προς την πληροφόρηση, δηλαδή αν, αν και υπάρχουν πληροφορίες που δεν πρέπει να δημοσιεύονται, θα πρέπει να ε, μπορεί να γίνεται αίτηση για παραχώρηση στοιχείων. Ζήλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ, αλλά ο συντονιστής αντικαθιστώ και τους ε, συναδέλφους. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Καπούτο για το σχέδιο γνωμοδότησης και όταν λέω εγώ θα εννοώ τον κύριο Τοσανόφσκι. Θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να βελτιωθεί. Στόχος έχει λοιπόν εδώ πέρα στόχο έχουμε να δημιουργηθούμε στόχο έχουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα καταγραφής ε, των εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα για βαρέα οχήματα, φορτηγά και λεωφορεία θα δημιουργηθούν ε, νέες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις θα εξασθενήσει η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαίων κατασκευαστών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το ότι ο εισηγητής προσπαθεί εδώ πέρα να μειώσει το πεδίο εφαρμογή. Οι κατασκευαστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση δεν θα έχουν αυτές τις υποχρεώσεις ε, και δεν θα δημοσιεύουν τα δεδομένα εάν δεν εξάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αντιπαραγωγικό. Βλέπουμε συχνά επίσης πώς ε, αλλάζουν ε, στις εκθέσεις οι εφαρμοστικές διατάξεις, πράξη κατεξιοδότηση, κάτι με το οποίο είμαι αντίθετος επίσης μιλάμε για ε, έναν κανονισμό, οπότε έχουμε ρυθμιστικές απαιτήσεις που βασίζονται σε έλλειπη Πρέπει να περιμένουμε, θεωρώ τουλάχιστον, μέχρι το 2021, όταν θα έχουμε τα σχετικά δεδομένα από ένα κεντρικό αρχείο. Οπότε ο κύριος Τάσανες και αναμένει και την συνεργασία με τους συναδέλφους στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κιλόνεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι. Σας ενημερώνω ότι η Καταρίνα δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ και θα διαβάσω το μήνυμά της. Συνάδελφοι, καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές διοξυδίου του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων από τα νέα βαρέα οχήματα, τα δεδομένα για τα πρόσφατα εξουσιοδοτημένα φορτηγά θα πρέπει να καταγράφονται με ε, εναρμονισμένο τρόπο και κάποια θα είναι και δημοσίως διαθέσιμα. Υπάρχει ανάγκη να, υπάρχει μεγαλύτερη, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια για τον τομέα των μεταφορών ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των διαφορών παραγωγών. Θα πρέπει τώρα να συζητήσουμε εάν η συμμόρφωση ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα θα πρέπει να ε, είναι προσβάσιμη σε τρίτα μέρη και να χρησιμοποιείται για την παραγωγή. Επίσης για τις νέες δοκιμές για τα νέα βαρέα οχήματα θα πρέπει να σκεφτούμε εάν αυτά τα τεστ μελλοντικά θα αντέξουν στις νέες συνθήκες. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νταλούντε. Θέλετε το λόγο. Όπως βλέπετε ούτε ο κ. Μπακαντότη είναι εδώ, οπότε δυστυχώς ε, δεν θα έχετε κάποια συγκεκριμένα σχόλια από τους πράσινους. Θα μπορούσα να κάνω και εγώ κάποια γενικά σχόλια, αυτά τα οποία λέμε συνήθως οι πράσινοι, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα. Θα σας απαλλάξω από αυτό το βάρος. Σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Άλεξ Πάκου. Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα να πω πως καλοδεχούμενη η συζήτηση αυτή. Όπως είπαμε, οι εκπομπές ε, των βαρέων οχημάτων είναι το 1 τέταρτο των οδικών μεταφορών και θα αυξηθούν στο μέλλον αν δεν γίνει κάτι. Γι' αυτό η Κομισιόν στο πρώτο πακέτο κινητικόταση είπε ότι θα λάβει κάποια μέτρα για να μειώσει τις εκπομπές από αυτά τα βαρέα οχήματα αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι το πρώτο στοιχείο, το πρώτο νομοθέτημα για το θέμα αυτό και κοιτάζουμε ακριβώς την παρακολούθηση των εκπομπών. Ξεκινάμε από τους εύκολους στόχους και έτσι δεν θα έρθει διαφάνεια στην αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε το τι γίνεται με την κατανάλωση ε, καυσίμων των φορτηγών. Και θα ξέρουν βεβαίως ε, και οι εταιρείες ε, το τι καταναλώνουν τα οχήματα και μην ξεχνάμε ότι τα καύσιμα είναι το 1 τέταρτο του λειτουργικού κόστους αυτών των εταιριών. Επίσης θα ανοίξει η αγορά, θα υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα θέματα του πια, δεδομένα θα πρέπει να είναι δημόσια. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή βρίσκει την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης διαφάνειας στην αγορά αλλά και το, ε, της εμπιστευτικότητας κάποιων πληροφοριών για λόγους ανταγωνισμού. Λοιπόν, πρόκειται για το πρώτο βήμα. Τώρα η Κομισιόν εξετάζει και παδιαγραφές εκπομπών για τα βαρέα οχήματα, για το διοξίδιο του άνθρακα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Δίνω ξανά τον λόγο στον κύριο Καπούτο. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους. Ε, χαίρομαι που συμφωνούμε στις βασικές αρχές ε, και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή δουλειά στον τομέα αυτόν γιατί θεωρώ ότι η κοινωνία απαιτεί όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια και πρέπει και εμείς να είμαστε κάπως πιο φιλόδοξοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Καπούτο. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι 18 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Αυτά. Και τώρα. Συνεχίζουμε και κλεισμένων των θυρών. Ένα σύντομο διάλειμμα και διακοπή του web streaming, πάδι, ώστε να μπορέσει και το κοινό να φύγει από την αίθουσα. Όσοι μπορούν να μείνουν είναι εκείνοι που είναι ε, υπεύθυνοι για σημαντικά ντοσχέ και που πρέπει να μας ενημερώσουν για τις διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε σύντομα και όσοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις μείνετε εντός της αιθούσης.